Dear colleagues, uh, eh, senior Commissario, dear Commissioner. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί επιτρόποι, σήμερα δεν είναι μόνο η τελευταία μας συνεδρίαση πριν από τις ενέργειες αλλά είναι το τελευταίο τμήμα της ε, συνεδρίασης που ξεκίνησε από εχθές. Ε, είχαμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη και συνεχίζω στα Ιταλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επιτρόπο για την ε, παρουσία του εδώ. Είχαμε την ευκαιρία να τον συναντήσουμε ήδη δύο φορές με την αρχική ακροαματική διαδικασία πριν από δύο μήνες. Σας ευχαριστούμε για την ε, διαθεσιμότητά σας. Εμείς ως Επιτροπή έχουμε κάποιες αρμοδιότητες που αφορούν στο χαρτοφυλάκιό σας και προσβλέπουμε συνέχιση αυτού του διαλόγου με την Κομισιόν. Σε σχέση με την προηγούμενη φορά λοιπόν έχουμε κάποιες καινοτομίε της στρατηγικής Digital Single Market το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα για διάφορους λόγους και σκέπτομαι τα πνευματικά δικαιώματα αλλά και την πρόσβαση στο περιεχόμενο του οπτικού ακουστικού μέσου, την προστασία των αλήκων, του ψηφιακού υλικού και η παραγωγή του υλικού που είναι ένα μεγάλο στίχημα για την Ευρώπη αλλά εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για την πρόοδο της ε, επανεξέτασης της ε, οδηγίας ε, BMS Είχαμε και στην προηγούμενη εντολή εκθέσει της Κομισιόν επ' αυτού που απέναντι στην αυξανόμενη σύγκληση και στην ανάγκη του να έχουμε ένα ισότιμο παιχνίδι απέναντι σε όλους τους φορείς του οπτικού ακουστικού υλικού. Χρειαζόμασταν μια ενδελεχή επανεξέταση της οδηγίας. Ε, γνωρίζουμε ότι εκκίνησε μια διαβούλευση, μια διαδικασία διαβουλεύσεως για την εφαρμογή της οδηγίας σε όλες τις χώρες. Ελπίζουμε ότι αυτή θα ολοκληρωθεί εντός της ε, προθεσμίας ώστε να παρουσιαστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχεδίου Juncker ώστε στους πρώτους μήνες του 2016 να είμαστε θέση να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Επίσης μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το ίδιο πρόγραμμα επενδύσεων ε, του σχεδίου Juncker να συμπεριλαμβάνει μία πτυχή και μία σημαντική προσοχή στις υποδομές, ε, τους ψηφιακούς αυτοκινητοδρόμους όπως ονομάζονται, που θα είναι ένα άλμα ποιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της ε, απαιτούμενης ανταγωνιστικότητας, αλλά και στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης προσοχής τις νέες αρμοδιότητες μας σχετικά με την ηλεκτρονική εκμάθηση και εκπαίδευση, επί των οποίων ε, ήμασταν σε επαφή με τις ε, Γενικές Διευθύνσεις ε, και τις αρμόδιες υπηρεσίες κομισιών και την ευρυζωνική κάλεψη των σχολικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μας ενδιαφέρει πολύ και το θέμα του Προπολογισμού Μάλιστα το κοιτούμε με μια κάποια ανησυχία ε, σχετικά με τις ε, περικοπές αυτές που έχουν ανακοινωθεί μεσοπρόθεσμα και στο EuroMed που είναι πολύ σημαντικό θέμα για μας. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια επί των οποίων υπάρχει μια ανάγκη εμβάθυνσης. Θα δώσω, σας δώσω αμέσως το λόγο για 10 λεπτά θα έλεγα περίπου για μια παρουσίαση και μετά θα έδινα το λόγο στους ε, συντονιστές ίσως τρία λεπτά για τον καθένα, για να δούμε ποιες άλλες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις θα μπορούσαμε να έχουμε. Ε, ευχαριστούμε εκ νέου για την παρουσία σας. Έχετε το λόγο, Επίτροπε. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητές κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, νέα πρόσκληση που μου κάνατε σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω για ορισμένα θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν. Είμαι εδώ για να απαντήσω στις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας σχετικά με το τι έχει γίνει στο παρελθόν, τι εμπειρίες έχουμε αποκομίσει, τι έχουμε κάνει μετά από τα τελευταία σχόλιά σας την προηγούμενη φορά που βρέθηκα εδώ. Πριν από λίγες μέρες έλαβαν χώρα οι διαβουλεύσεις σχετικά με την οδηγία για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Συζητήθηκε το πώς οι φορείς της αγοράς βλέπουν την κατάσταση και ποια είναι τα Επόμενα βήματα, πρώτον σχετικά με την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα, όπου σκοπεύουμε να χτίσουμε πάνω στην πράσινη βίβλο που δημιουργήθηκε πριν από δύο χρόνια, καθώς επίσης και να συνεχίσουμε βασισμένοι στις ε, εκθέσεις της ε, κυρίας Καμερέβερτ και της Επιτροπής σας, ε, όπου εντοπίστηκε ανάγκη επανεξέταση της υφιστάμενης κατάστασης. Οι υφιστάμενες ρυθμίσεις είναι από το 2007. Είναι λοιπόν κάπως παλιές και χρειάζονται αναθεώρηση και επικαιροποίηση. Έτσι ώστε μέσα στο 2015 να έχουν ολοκληρωθεί, να έχει ολοκληρωθεί αυτή η επαναξιολόγηση στα πλαίσια του κανονισμού refit, να εξεταστούν οι επιλογές που έχουμε έτσι ώστε να εξελιχθεί και να επικαιροποιηθεί περαιτέρω ο κανονισμός. Μετά από τις αναλύσεις μας καταλήξαμε σε μία περιεκτική εικόνα της κατάστασης και σκοπεύουμε τα επόμενα χρόνια, μετά φυσικά από διαβουλεύσεις με εσάς, να παρουσιάσουμε την επικαιροποιημένη οδηγία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. πρέπει να ασχοληθούμε καταρχάς με το εξής ε, ερώτημα. Εάν χρειάζονται επικαιροποίηση και επαναξέταση όλοι οι φυστάμενοι κανόνες. Έπειτα, πρέπει να δούμε εάν χρειάζεται μια κλιμακωτή ρύθμιση, ένα κλιμακωτό σύστημα όπως μέχρι τώρα, και εάν χρειάζεται να αλλάξουμε τις υφιστάμενες δομές. Ε, χρειάζεται να εξετάσουμε την προστασία των ανηλίκων, την προστασία των ευρωπαϊκών πολιτισμικών αγαθών, τον περιορισμό της διαφήμισης ή την απαγόρευση της διαφήμισης, τον τηλεοπτικό δηλαδή ραδιοφωνικό χρόνο που θα επιτρέπεται να έχουν οι διαφημίσεις και το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Ε, να σας αναφέρω χαρακτηριστικά τις διαφημίσεις για τον καπνό και το αλκοόλ. Είναι αναγκαία λοιπόν αυτή η αναθεώρηση στους τομείς αυτούς. Πρέπει να δούμε αν χρειάζεται αλλαγή ή κατάργηση. Επίσης, χρειάζεται μία αξιολόγηση της σχέσης με τους ε, τηλεοπτικούς φορείς, με τις ε, δημόσιες ε, και ιδιωτικές συνεργασίες, συνεργασίες δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Η προσβασιμότητα αυτών στους πολίτες Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια σχετική ρύθμιση στον εγγονισμό για τα οπτικοακουστικά μέσα. Υπάρχουν όμως άλλους κανονισμούς, άλλες οδηγίες. Επίσης, πρέπει να εξεταστεί το ερώτημα των ίσων όρων ανταγωνισμού. Να δούμε τι περιλαμβάνεται στην οδηγία σχετικά με τους ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους ενδιαφερόμενους εδώ παρατηρήσαμε την ε, ανάγκη μερικών αλλαγών ε, μιας επέκτασης του πεδίου εφαρμογή. που να περιλαμβάνει την προστασία των ανηλίκων, το κοινό συμφέρον, συγκεκριμένες ε, απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, επιτροπές εποπτείας και ελέγχου των διάφορων επιμέρους ομάδων, Είναι αναγκαίες όλες αυτές οι ενέργειες, όμως δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν σε όλες ε, τις ε, πτυχές της οδηγίας. Πρέπει να αναρωτηθούμε τι χρειάζεται, τι είναι τεχνικά δυνατό, έτσι ώστε να δημιουργηθούν πραγματικά αυτοί οι ίσοι όροι ανταγωνισμού και να αλλάξει το τοπίο σε σχέση με τα δέκα τελευταία χρόνια. Είμαι έτοιμος να συζητήσω μαζί σας στη διάρκεια του έτους ε, σχετικά με τον κανονικό, κανονισμό Refit. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι ο τομέας ε, των ψηφιακών μέσων, των ε, ραδιοτηλεοπτικών μέσων, είναι ένας τομέας που χαρακτηρίζεται από ταχύτατες αλλαγές. Τόσο γρήγορες μάλιστα που δεν προλαβαίνουμε να εφαρμόσουμε την νέα νομοθεσία γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Θέλουμε ε, δύο-τρία χρόνια μέχρι να εφαρμόσουμε στην εθνική νομοθεσία τα νέα δεδομένα. Μέχρι τότε έχουν αλλάξει όμως. Έχει αλλάξει το τοπίο. Μένουμε πίσω και χάνουμε σε αξιοπιστία. Και αυτή η ενέργεια είναι μια αναστρέψιμη. Και θα ήθελα λοιπόν να θέσω το ερώτημα ενώπιον της Επιτροπής σας, αν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο γρήγοροι στην επεξεργασία μας, μαζί με το Συμβούλιο, έτσι ώστε μέσα στο 2006 να άρουμε όλους τους ε, φραγμούς που οδηγούν σε καθυστερήσεις, έτσι ώστε το Συμβούλιο να είναι τόσο γρήγορο όσο και εσείς, για να μπορεί να εφαρμόσει το γρηγορότερο δυνατόν την αναθεωρημένη οδηγία. Χρειαζόμαστε λοιπόν ενδελέχεια, ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Επιπλέον, Σίγουρα το πιο δύσκολο κομμάτι του έργου μας είναι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ψηφιακό χώρο. Και εδώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μου επισημάνατε κάποια πάρα πολύ σημαντικά και κέρια θέματα σχετικά με αυτό. Επεξεργασία, τυποποίηση και χρήση των ψηφιακών μέσων, ανεξάρτητα αν μιλάμε για μουσική, για κάποιο βιβλίο, για μια εφημερίδα, για ταινία που είναι σε, ψηφιακό, σε ψηφιακή μορφή η ψηφιακή τεχνολογία πλέον έχει εξαπλωθεί και περιλαμβάνει τα πάντα. Και πιστεύω πως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν στα δικαιώματα μάλλον πνευματικής ιδιοκτησίας δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο οι τεχνικές λεπτομέρειες αλλά και η πολιτική διάσταση. Ο δημιουργός, είτε είναι συγγραφέας, είτε είναι συνθέτης, είτε είναι σκηνοθέτης, ή δημοσιογράφος, μουσικός, έχει δικαιώματα και πρέπει να του δώσουμε μια προοπτική έτσι ώστε να μπορεί να απολαμβάνει των δικαιωμάτων του. Αναφερόμαστε πολύ συχνά στα δικαιώματα πνευματικής ε, ιδιοκτησίας και στο copyright, λες και είναι το ίδιο πράγμα. Είναι όμως διαφορετικά. Άλλα τα δικαιώματα του δημιουργού και άλλα τα δικαιώματα της πνευματική ιδιοκτησίας. Χρειάζεται λοιπόν διαφορετική αφετηρία για το καθένα. Και αυτό κατέστησε αφές την περασμένη Πέμπτη στο Στρασβούργο, στη σχετική συζήτηση. Ωστόσο πιστεύω πως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται αυτή την στιγμή και να κάνουμε πράξεις. Η πολιτική δεν είναι μόνο λόγια, είναι και εφαρμογή. Πρέπει να νομοθετήσουμε λοιπόν έτσι, ώστε η τεχνολογία να μην μας ορίζει. Και εδώ να πω ότι η πνευματική εργασία είναι κάτι που θα πρέπει να έχει μέλλον. Πρέπει να δώσουμε μια προοπτική για το 15χρονο που θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική, με τη δημοσιογραφία, με κάποιο άλλο δημιουργικό επάγγελμα. Πρέπει να του δώσουμε ασφάλεια και βεβαιότητα ότι θα μπορέσει να ζήσει από αυτό επαγγελματικά. Ως χρήστες, επίσης, διαβάζουμε εφημερίδες, ακούμε μουσική, βλέπουμε κινηματογραφικές ταινίες. Όλοι λοιπόν και οι χρήστες έχουμε συμφέρον να συνεχίσουν να βγαίνουν νέα προϊόντα τα οποία θα είναι άμεσα προσβάσιμα. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε την σωστή ισορροπία ανάμεσα στο χρήστη και στην διαδικτυακή κοινότητα, την ψηφιακή κοινότητα, την κοινότητα της ε, πληροφορίας και της εκπαίδευσης και από την άλλη στους δημιουργούς οι οποίοι θα δίνουν τον κόπο τους για τον χρήστη. Επίσης πρέπει να μιλήσουμε για θεμελιώδεις αρχές, όπως την φορητότητα για παράδειγμα, να έχουν όλοι στην Ευρώπη τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα πνευματικά έργα χωρίς περιορισμούς. Αυτή είναι μία αρχή. Η αρχή της διασυνοριακής πρόσβασης για τους καταναλωτές. Αυτές οι αρχές όμως για μένα δεν είναι θέσφατα. Είναι αρχές που χωρούν και εξαιρέσει. Και εδώ να αναφέρω τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. ο οποίος χαρακτηρίζεται από την πολυμορφία, από την πολυμορφία εξαιτίας των διαφορετικών γλωσσών, των διαφορετικών πολιτισμών. Και χρειάζεται να δώσουμε ένα μέλλον, μια προοπτική για το μέλλον στον κλάδο αυτό. Ο αθλητισμός επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Χρειάζεται να υπάρχει μια προοπτική χρηματοδότησης και να μην γίνονται εξαιρέσει ανάμεσα σε αθλήματα πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Επίση, πρέπει να μιλήσουμε για εξαιρέσει, για συγκεκριμένε ομάδες εξαιρέσεων. Για παράδειγμα, τα πνευματικά δικαιώματα και τους ε, ανθρώπου με αναπηρία. Οι άνθρωποι με αναπηρία πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση η κατάρτιση επίσης, και εκεί υπάρχουν εξαιρέσεις για ορισμένες ε, εγκαταστάσεις όπως βιβλιοθήκες που φιλοξενούν πολιτισμό. Επίσης, στον χώρο της έρευνας πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται εξέταση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι κανόνες δεν πρέπει να περιορίζουν. Το αντίθετο, πρέπει να δίνουν δυνατότητες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις εξαιρέσεις αυτές έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι πολίτες. Επίσης, σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε την πρότασή μας για τα πνευματικά δικαιώματα μέχρι το τέλος του 2015. Επίσης, ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών μας. Είναι το τρίτο θέμα που θέλω να σας ε, παρουσιάσω σήμερα. Ο μεγάλος ε, συνασπισμός των ψηφιακών μέσων επεκτείνεται. Έχουμε δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσει εργασίας στον τομέα της, πληροφορική, ε, και σκοπεύουμε κάθε χρόνο να αυξάνουμε τις νέες θέσει απασχόλησης, να αυξάνουμε τους ε, φορείς που θα συμμετέχουν, που θα δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης στον τομέα της πληροφορικής. Και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν έχουμε αρκετές θέσεις σπουδών για τον κλάδο αυτό. Εάν θέλουμε να γίνουμε κι εμείς μια δεύτερη Silicon Valley, πρέπει να δώσουμε τις κατάλληλες βάσεις γι' αυτό. Και αυτή η αξία πρέπει να δημιουργηθεί εδώ, έτσι ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο για να δημιουργηθούν και οι δεξιότητες που χρειάζονται. Και είναι ευθύνη μας να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι χρειάζεται, χρειάζονται νέες, νέα μυαλά, νέοι επιστήμονες στον χώρο της πληροφορικής. Επίσης, όσον αφορά τις ε, συχνότητες, τις ε, συχνότητες ε, MHz στους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Χρειάζεται βελτίωση των τηλεπικοινωνιών. Πρέπει όμως να προσέξουμε να μην βελτιώσουμε έναν τομέα και επιδεινώσουμε κάποιον άλλο. Να μην υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στις ε, τηλεπικοινωνίες και στην ραδιοτηλεόραση. Αυτή τη στιγμή το επιτελείο μου προετοιμάζεται για την ε, διάσκεψη στη Γενέβη τον Νοέμβριο και η προετοιμασία που πρέπει να κάνουμε πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή. Χρειαζόμαστε λοιπόν την συνδρομή όλων σχετικά με πολλούς τομείς όπως η ευρυζωνικότητα, η ψηφιακή ευρυζωνικότητα. Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν οδικό χάρτη, ο οποίος να εφαρμοστεί ταυτόχρονα από όλα τα κρατημέλη. Και πιστεύω πως η έκθεση του κυρίου Λαμέ είναι μια πάρα πολύ καλή βάση για να προετοιμαστούμε. Τέλος, Euronet. Χρειάζεται περισσότερη... Χρειάζεται περισσότερη ραδιοτηλεοπτική φορή. Euronet Euronews. Χρειαζόμαστε σωστά θεμέλια. στους ε, ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν με όσο το δυνατόν οικονομικότερο κόστος ώστε να προσφέρουν εξίσου ποιοτικό περιεχόμενο παντού. Επίσης, συμφωνώ με σας για την δημιουργία σταθερής χρηματοδότησης σχετικά με, για το Euronet. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό επανδρομένο από καταρτισμένο προσωπικό. Είχα πολύ επικοδομητικές συνομιλίες με τον διευθυντή του Euronews στη Λιόν πρόσφατα και συζητήσαμε τα προβλήματα, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Euronews και ο, τα προβλήματα αναζήτησης εταίρων και την ανάγκη επενδύσεων που, που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η κακή πορεία του Euronews, ιδιαίτερα σε σχέση με τον ανταγωνισμό που προέρχεται από τις τρίτες χώρες, από τη Ρωσία για παράδειγμα. Όπως ε, ξέρετε, το Euronews δεν είναι ευρωπαϊκός οργανισμός. Ε, στηρίζεται από ευρωπαϊκά κονδύλια, όμως μέτοχοι του Euronews είναι τα κράτη-μέλη. Διεξάγαμε συνομιλίες με τους ε, ενδιαφερόμενους ε, φορείς, ενδιαφερόμενους μετόχους, ε, συγκεκριμένα τον κύριο ενδιαφερόμενο από την Αίγυπτο. Και μπορώ να σας πω ότι οι συνομιλίες ήταν αρκετά επιτυχείς, ήταν αρκετά θετικές στηρίχθηκε η πρόταση του από την γαλλική και ιταλική ραδιοτηλεόραση και συζητήθηκε το ενδεχόμενο πώληση ενός μερίδιου στον επενδυτή αυτών. Έπειτα δημιουργήθηκε ένα ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο το οποίο μπορεί να αναλάβει καθήκοντα μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα σχετικά με τον έλεγχο. Έλεγχο περιεχομένου του προγράμματος και την αντικειμενική απεικόνηση των ε, κρατών. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μία ανάλυση για να διαπιστώσουμε πού έχουν σημειωθεί συγκρούσεις ε, με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και πού υπάρχουν μεροληπτικές απεικονίσεις. Εν ώψη του 2016 θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε και το Euronet και το Euronews να έχουν επαρκή χρηματοδότηση διότι πρέπει να αποφύγουμε να επιλέξουμε ένα από τα δύο, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και ε, τα δύο ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση. Μας είπε πολλά επίκαιρα στοιχεία σχετικά με την οδηγία DNS για τους στόχους του 16 και για την ε, συμπλήρωση της όλης διαδικασίας με ένα κάποιο follow-up το οποίο μας ενδιαφέρει εφόσον έχουμε ξεκινήσει να συζητούμε από αυτού από την αρχή εμείς. Τώρα για το Euronet και το Euronews και τα λοιπά εμείς μόλις σήμερα ε, εγκρίναμε τις τροπολογίες για τις γνωμοδοτήσεις του προϋπολογισμού και είχαμε και μια συγκεκριμένη επί του, επί του Euronet και ένα αίτημα αύξησης των σχετικών προβλέψεων του προλογισμού γιατί είδαμε και περικοπές. Θα ζητούσαμε λοιπόν μια δέσμευση ισχυρή από την Κομισιόν ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια γραμμή της μη μείωσης των χρηματοδοτήσεων για αυτά τα θέματα έτσι όπως είχαν προβλεφθεί. Ε, τώρα διάφορες συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο για παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Παρακαλώ με τη σειρά που τους εγγράψαμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που για άλλη μια φορά είστε παρόν στην Επιτροπή μας με πραγματικά εντατικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων πολύ σημαντικό για τον τομέα της δημιουργίας, τον πολιτισμό Έχουμε θέματα στην ημερήσια διάταξη που σαφώς ε, θα μας επιτρέψουν να συντονίσουμε την δράση μας. Βεβαίως ε, υπάρχουν πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα και τα οποία θα πρέπει να εξισορροπήσουμε με δίκαιο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που ε, είστε σήμερα εδώ. Καταρχήν το θέμα της οδηγίας για τα ακουστικά μέσα. Σας ευχαριστώ γιατί πραγματικά η ταχύτατη αντίδρασή σας είναι κάτι που μας επιτρέπει και εμάς να μην περιμένουμε πολύ μέχρι να μπορέσουμε να γνωμοδοτήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιδρούμε με ταχύτητα σε αυτά τα θέματα καθότι η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτητα και θα πρέπει να μπορούμε με συντομία να επιλύουμε θέματα που προκύπτουν έτσι ώστε να μην εμποδίζουμε την υλοποίηση και την εφαρμογή ε, αυτών των κανονισμών. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω γιατί οι διαβουλεύσεις ξεκίνησαν ταχύτητα, έχουν εντοπιστεί οι δυσκολίες και εμείς ε, βεβαίως έχουμε έγγραφα και στοιχεία. Η ερώτησή μου είναι μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτή η διαβούλευση και πότε θεωρείτε θα έχετε μια πρώτη εκτίμηση. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι από την αρχή του 2016 μέχρι τα, ε, τους πρώτους μήνες, μέχρι την Άνοιξη, να ανταποκριθούμε και να έχουμε ολοκληρώσει την δική μας ε, τοποθέτηση. Τώρα όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, το copyright, τα λεγόμενα δικαιώματα δημιουργών, Είναι πολύ σημαντικό εδώ οι χρήστες, οι καταναλωτές, αυτοί οι οποίοι θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, να ληφθούν υπόψη αυτοί και τα δικαιώματά τους. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και οι ενδιάμεσοι, αυτοί οι οποίοι παρέχουν την ε, υπηρεσία. Δεν είναι δηλαδή σημαντικό μόνο να δούμε αυτόν που δημιουργεί και αυτόν που καταναλώνει τελικά το ε, έργο τέχνης, το προϊόν της δημιουργίας, αλλά και όλη η ενδιάμεση. Ο συγγραφέας ή ο δημιουργός, είτε πρόκειται για δημοσιογράφο ή για κάποιον ο οποίος δημιουργεί, δεν είναι πάντα σε θέση να διαπιστώσει όλες τις ιδιαιτερότητες ε, της αγοράς, τα δίκτυα από τα οποία πρέπει να περάσει. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε πού χρειάζονται προσαρμογές, πού οι ενδιάμεσες δομές και τα δίκτυα μπορούν να παίξουν ένα ρόλο θετικό έτσι ώστε η διάθεση στην αγορά να ληφθεί υπόψη το θέμα των εκδοτών, το θέμα αυτών που αναμεταδίδουν αυτά τα έργα και τα δικαιώματα τα οποία άπτονται όλων αυτών των ενδιάμεσων δομών. Οι εξαιρεσει είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι βεβαίως πρέπει να παραμείνουν εξαιρέσεις και να μην γίνουν κανόνες. Στο θέμα της έρευνας πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τι είναι απαραίτητο, τι χρειάζεται εδώ να στηρίξουμε και να προωθήσουμε και να σκεφτούμε ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των εξαιρέσεων. Μέχρι ποιο βαθμό θα τις προστατεύσουμε και θα τις δεχτούμε παραδείγματος χάρη το θέμα του τομέα της εκπαίδευσης. Αυτός σαφώ και θα πρέπει να ε, εξαιρεθεί για τον τομέα της παιδείας. Υπάρχει εξαίρεση και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει αυτό να συνεχιστεί. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών βιβλίων, των εγχειριδίων, μέχρι πού όμως μπορεί η αναμετάδοσή τους να γίνεται χωρίς ε, επιβάρυνση. Και εδώ χρειάζεται ισορροπημένη προσέγγιση το θέμα της έρευνας και της στήριξης των εταιρικών σχέσεων μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα πιστεύω ότι για τα πανεπιστήμια και τη σχέση τους, τη συνεργασία τους με επιχειρήσεις επίσης, η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και η δυνατότητα να μην επιβαρύνονται με δικαιώματα τα δημιουργήματα αυτά τα οποία έχουν σαν σκοπό την χρήση τους σε περιβάλλοντα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Συμφωνώ επίσης και με τις προτάσεις σας όσον αφορά το ραδιοφωνικό δίκτυο, αλλά θα πρέπει εδώ να δούμε λίγο και τους μικρούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, τους τοπικούς, περιφερειακούς, και όχι μόνο τους μεγάλους ε, ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα μεγάλα εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, γιατί είναι εξίσου σημαντικό να στηρίξουμε και την τοπική ε, ραδιοφωνική αναμετάδοση, η οποία πολλές φορές μπορεί να εμπλουτίσει το περιεχόμενό της και με ευρωπαϊκό περιεχόμενο, ευρωπαϊκές ειδήσει. Για το Euronews δεν είμαι τόσο ευτυχής με αυτά που συμβαίνουν Ξέρουμε με την υπόθεση της Ουκρανίας και της Ρωσίας τι συνέβη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τη διαφάνεια. Η Ουκρανία είναι ένα παράδειγμα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, αλλά είναι πολύ κρίμα αν οι ειδήσει αναμεταδίδονται με μη αντικειμενικό τρόπο όπως από ό,τι φαίνεται συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Και θα πρέπει εδώ κάτι να γίνει με το Euronews. Χαίρομαι που το Συμβούλιο έχει πάρει αυτές τις αποφάσεις, αλλά είναι συγκεκριμένο να δούμε ποιες είναι οι ομάδες, οι κοινότητες και τα συμφέροντα που τελικά προωθούνται και εκπροσωπούνται για να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει αντικειμενικότητα και με μεγάλη χαρά θα σας πρότεινα αυτός ο διάλογος που έχουμε ξεκινήσει να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κάμερβερτ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τίγκερ, που είστε σήμερα εδώ. Όλα αυτά τα θέματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα μας τα παρουσιάσετε και διατυπώσατε και τις σωστές ερωτήσεις. Ανυπομονούμε να δούμε εξάλλου και ποιες θα είναι οι απαντήσεις της Επιτροπές για αυτά τα τόσο σωστά ερωτήματα. Αναφερθήκατε στα οπτικοακουστικά μέσα, στην οδηγία, στο θέμα της ευθύνης του φορέα παροχής υπηρεσιών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών υπεύθυνο για το περιεχόμενο. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για αυτό το σημείο. Φοβάμαι ότι θα πέσουμε στην παγίδα του ελέγχου του περιεχομένου, κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε αυτό το επίπεδο. Το θέμα της προστασίας των νέων τώρα. Και εδώ υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το θέμα της προστασίας. Ξέρετε ότι και η εκτίμηση είναι τελείως διαφορετική. Υπάρχουν ταινίε που επιτρέπονται, είναι κατάλληλες για παιδιά 12 ετών στη Μεγάλη Βρετανία και απαγορεύονται στην Γερμανία. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε ποια είναι τα πρότυπα που μπορεί ενδεχομένως να εφαρμοστούν Στη Γερμανία ο τρόπος ε, προστασίας βασίζεται στην αυτορύθμιση. Είναι κάτι που έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά μέχρι τώρα και το ίδιο θα έλεγα συμβαίνει και ισχύει και για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν παρεμβαίνει το Υπουργείο ή οι εθνικές αρχές για να αποφασίσουν αν είναι κατάλληλο ή ακατάλληλο και από ποια ηλικία επιτρέπεται ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Η αυτορύθμιση λοιπόν λειτουργεί ικανοποιητικά. Σκεφτείτε το και αυτό. Τα σημαντικά σημεία της παρουσίασής σας νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα το θέμα των ε, πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων του δημιουργού, το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας ε, κάποιων έργων τέχνης και πρέπει να βρούμε ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των δικαιωμάτων, των χριστών αλλά βεβαίως και των δημιουργών που δεν μπορούμε να μην τα προστατεύσουμε με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Νομίζω ότι το πολιτιστικό περιεχόμενο που φτάνει τελικά μέχρι τον τηλεθεατή, μέχρι τον Ευρωπαίο πολίτη είναι σημαντικό. Κάτι που δεν φτάνει ποτέ σε αυτόν, καταλαβαίνετε ότι πλέον χάνει και το νόημά του. Εάν δηλαδή οι δομές είναι τόσο περίπλοκες που η πρόσβαση σε ένα πολιτιστικό αγαθό είναι εξαιρετικά δύσκολη, χάνουμε την ουσία. Θα ήθελα επίσης να πω ότι τις τελευταίες ημέρες εκνευρίστηκα λίγο από τις δηλώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ουδετερότητα των δικτύων και τις διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει με την Επιτροπή. Βεβαίω ε, δεν έχουμε εντολή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Ούτε μπορούμε να απαγορεύσουμε ε, κάτι και φυσικά και δεν έχουμε πάρει και καμία τελική απόφαση. Αλλά συζητήσαμε το θέμα και στον τελικό κύκλο, αν θέλετε, των διαπραγματεύσεων Συζητήσαμε και την θέση και τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ουδετερότητα των δικτύων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να διαπιστώσουμε ότι στο θέμα αυτό αλλά και στις ευρυζωνικές Άδειε που δίνονται, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε ότι η τοποθέτηση της Επιτροπής μπορεί να γίνει δεκτή από εμάς. Πρόκειται για μια προσέγγιση που σίγουρα δημιουργεί στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι στις τηλεπικοινωνίες προσφέρουν συμβάσεις και συμβόλαια για την εταιρεία Netflix, για το Spotify, λέγοντας παραδείγματο χάρη ότι δεν μας ε, αφορά το τι θα γίνει με τον ε, ανταγωνισμό, ότι δεν μας αφορά η προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού και ότι θέλουμε σε κάθε περίπτωση να μην αμφισβητήσουμε τα πνευματικά δικαιώματα, σε αυτή την περίπτωση σίγουρα η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στη μουσική, στον κινηματογράφο κτλ. δεν μπορούν να διασφαλιστούν. Το λεγόμενο zero rating είναι κάτι που σημαίνει ότι και τα κινηματογραφικά ε, έργα αλλά και η μουσική, ιδιαίτερα για πιο μικρούς φορείς, δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να προστατεύονται. Αυτό που λέει εδώ η Επιτροπή το κατανοώ διότι ουσιαστικά προασπίζεται την ελευθερία, τον ανταγωνισμό. Αλλά θα πρέπει να δούμε γενικότερα το θέμα, το θέμα του γιουρανετόδα η χρηματοδότηση Πώς μπορούμε να τη διασφαλίσουμε. Για το Euronews εγώ ε, θα ήθελα να ασκήσω εντονότατη ε, κριτική. Δεν έχει σημασία αν χρηματοδοτείται ναι ή όχι από την Επιτροπή αυτός, ε, αυτή η επιχείρηση, αυτός ο σταθμός. Μέχρι τώρα ήμασταν πολύ θετικοί γιατί η παρουσίασή τους για τα ευρωπαϊκά θέματα ήταν ικανοποιητική. Το θέμα όμως είναι ότι όταν έρχεται σήμερα κάποιος αγοράζει ένας ε, ολιγάρχης θα έλεγα ξεκάθαρα αγοράζει κάποια δικαιώματα ενός τηλεοπτικού σταθμού για να έχει την ε, παρουσίαση των ειδήσεων όπως επιθυμεί, καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει παρέμβαση. Είτε πρόκειται για Ρώσο ολιγάρχη, είτε πρόκειται για Ουκρανό ολιγάρχη. Αυτό δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην χρηματοδότηση αυτού του σταθμού, από τη στιγμή δηλαδή που υπάρχει δημόσια κρατική χρηματοδότηση, ελπίζω να μπορούμε να διασφαλίσουμε και στο μέλλον την αντικειμενικότητα και τη σωστή παρουσίαση των γεγονότων από αυτό το σταθμό. Πραγματικά θα πρέπει να διατηρήσουμε ένα μοντέλο χρηματοδότησης ή συνχρηματοδότησης που να βασίζεται σε αυτά που συμβαίνουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία, όπως δηλαδή λειτουργούν και χρηματοδοτούνται οι ε, δημόσιοι, οι κρατικοί, τηλεοπτική και ε, ραδιοφωνική σταθμοί. και να υπάρχει μια ανεξαρτησία όσον αφορά ε, την γραμμή που ακολουθούν οι δημοσιογράφοι, γιατί αυτό είναι κάτι που πλήττει την αξιοπιστία της Ευρώπης. Ευχαριστούμε ο κύριος ε, Λίουερ, μετά Τρούπελ και μετά θα ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο γύρο για να έχουμε κάποιες απαντήσεις. Θα, θα παρακαλούσα όμως λέει η Πρόεδρος να μείνουμε στα τρία λεπτά αν μπορούμε. Ναι πρόεδρε θα προσπαθήσω, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο και εγώ θεωρώ ότι όταν πληρώνει κανείς για να μάθει νέα που είναι ένα αμφισβητήσιμο πρότυπο σε κάθε περίπτωση είναι ένα καλύτερο πλαίσιο από το πλαίσιο των ενισχύσεων ή των επιδοτήσεων. Ε, με προβληματίζουν κάπως αυτά που ακούω, τα σχόλια που ακούω σχετικά με το Euronews και είναι αξιοσημείωτο που συνάδελφοι από το S&D, ECR που εκφράζουν αντίστοιχες ανησυχίες και νομίζω ότι αυτό αξίζει κανείς να το παρατηρήσει καθεαυτό, την παρατήρηση δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το υβριδικό μοντέλο με επιδοτήσεις αλλά και ιδιωτική ιδιοκτησία, ε, συντακτικό έλεγχο κτλ. Όλο αυτό το μίξ δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Ένα ελεύθερο πρότυπο είναι πάντοτε καλύτερο από τη διαχείριση των ειδήσεων. Και αυτό δεν έχει καθόλου καλή δεν απεικονίζει με καθόλου καλό τρόπο ή θετικό τρόπο την Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν δημιουργούμε μια σύγχυση με αυτά τα υβριδικά πρότυπα επί του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, πέραν του αν είναι, πέραν του αν είναι χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος σε στιγμές σαν αυτές που διερχόμεθα. αντί για άλλα προγράμματα που θα μπορούσε να διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καθόλου να δαπανά. Επίσης, χρειάστηκαν εννέα εβδομάδες για να λάβω απάντηση στο ερώτημά μου που υπέβαλα για το Euronews και μετά κατά θαυμαστή σύμπτωση, όταν είπα ότι δεν είχα λάβει απάντηση, έλαβα εντός τριών ωρών. Απίστευτο δεν το βρίσκεται. Θα ήθελα λοιπόν αυτά να μην ε, συμβαίνουν είναι πολύ πιο εύκολο να απαντούμε σε μια ερώτηση παρά να βγαίνουμε στον τύπο και να λέμε ότι δεν είχαμε λάβει απάντηση. Έχω την εντύπωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τρούπε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Όταν για την παρουσίασή σας θα ε, αρχίσω από το τελευταίο σημείο που αναφέρατε. Καταρχάς ορίζω το γεγονός ότι αναφερθήκατε στην χρηματοδότηση του Euronet και να ξέρετε πως έχετε την επιτροπή μας με το μέρος σας. Θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με αυτό που είπε η Πέτρα Κάμερεβερ. Η συντακτική αναξαρτησία, η αναξαρτησία μάλλον των συντακτών είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να διασφαλιστεί και τίποτα άλλο δεν μπορούμε να ε, δεχτούμε. Πρέπει να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν θα είναι 100% ε, αναμειγμένη ή αν θα αποσυρθεί από το Euronet. Μία ενδιάμεση λύση, μία μεσοβέζικη λύση δεν μπορούμε να αποδεκτούμε. Έπειτα, μιλήσατε για την οδηγία τα οπτικοακουστικά μέσα. Και θεωρώ αποφασιστικές τις εξελίξεις για τις ε, συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Χρειάζεται μία ρύθμιση όπως είπατε και εσείς κλιμακωτή, πρέπει όμως να φροντίσουμε να διασφαλίζεται καλή πρόσβαση για όλους τους χρήστες και, ε, η... και χρειάζεται να διασφαλιστεί επίσης και η πρόσβαση σε ε, πολλούς φορείς. Επίσης, ε, θα αναφερθώ και εγώ σε κάτι που ανέφερε η κυρία Κάμερ Εβερτ. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ασκούμε έλεγχο επί του... Ε, ε, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να είναι υπεύθυνο ο πάροχος για το περιεχόμενο. Αυτό θα συνιστά παρέμβαση στις ε, υπηρεσίες που προσφέρουν αυτοί οι πάροχοι. Έπειτα, φορητότητα, φορητότητα περιεχομένου. Εάν για παράδειγμα μπορώ να συνεχίσω να έχω πρόσβαση στη συνδρομή μου σε μια διαφορετική χώρα ε, χαίρομαι πάρα πολύ που αναφερθήκατε σε αυτό, διότι πραγματικά αφορά την ε, πολιτισμική πολυμορφία. Χρειάζεται να βρούμε δυνατότητες ε, για την χρηματοδότηση επίσης του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Και εγώ θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ρωτήσω εσείς ποιες λύσεις βλέπετε, τι προτάσεις έχετε. Είναι σίγουρα ένα αρκετά επίμαχο ε, σημείο. Το, η δική μου πολιτική ομάδα έχει αντίθετη άποψη από εσάς. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια κατεύθυνση επιθυμείτε να ακολουθήσετε αυτή τη στιγμή, τι γίνεται ε, εκεί και αν θεωρείτε πως ε, η παρέμβαση είναι σωστή. Έπειτα, είδαμε πρόσφατα ότι, πραγμα... ότι είναι αρκετά αμφιλεγόμενο το θέμα των ε, φωτογρα... πανοραμικών φωτογραφιών. Σε ορισμένα κράτη-μέλη η πρόσβαση είναι ελεύθερη, σε κάποια άλλη υπάρχουν περιορισμοί για τα δικαιώματα των αρχιτεκτόνων που δημιούργησαν αυτά τα κτίρια κτλ. Εσείς τι προτάσεις έχετε σχετικά με το θέμα αυτό. Θα έλεγα να κλείσουμε αυτό τον πρώτο γύρο και θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο για τις απαντήσεις του. Κύριε Επίτροπε, ε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσες όλες τις ε, ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να τις απαντήσω όλες σήμερα, όμως σας υπόσχομαι ότι δεν προλάβω να σας ε, το απαντήσω γραπτό σε διεξοδικότερα στις ερχόμενες εβδομάδες. Όσον αφορά την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα, να σας πω ότι η φυστάμενη οδηγία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε γρήγοροι, διότι πρέπει να επιλύσουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, ε, τους ίσους όρους ανταγωνισμού, την είσοδο όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων και παρόχων για να εξασφαλιστεί αυτή η ισότητα του ανταγωνισμού. Επίσης, γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής, προστασία των καταναλωτών, τις ε, υπηρεσίες on demand. Χρειάζεται αναθεώρηση όλων αυτών και επίσης ε, να εξεταστούν τα ε, να εξεταστεί το περιεχόμενο που προκαλεί διακρίσεις, που υποκινεί μίσος. Αυτά είναι προβλήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία δέκα χρόνια, που πριν ήταν άγνωστα ή μικρότερη κλίμακα. Επίση, όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων, ε, να κάνουμε έναν διαχωρισμό ανάμεσα στη ραδιοτηλεόραση και στο video on demand. Πρέπει να δούμε εάν εκεί οι ρυθμίσεις είναι δίκαιες, εάν χρειάζεται να τις αλλάξουμε. Μετά πρέπει επίσης να δούμε πόσο αποτελεσματική είναι η νομοθεσία. Να δούμε εάν ο νομοθέτης με το έργο του επιτυγχάνει το στόχο που είχε θέσει πριν από 9 χρόνια, εάν οι στόχοι που είχαμε πριν από 9 χρόνια είναι ακόμα επίκαιροι, Επίσης, χρειάζεται να εξετάσουμε το θέμα του κόστους. Πρέπει να υπάρχει μία αναλογική σχέση κόστους χωρίς ε, υπερβολική γραφειοκρατία. και επίσης να απαντήσουμε στα ερωτήματα σχετικά με την έννοια αγορά. Μήπως οι εξελίξεις στον χώρο της αγοράς ε, δημιουργούν νέα δεδομένα τα οποία έρχονται σε αντίφαση με την υφιστάμενη νομοθεσία. Πού έχουν εντοπιστεί στην πράξη προβλήματα, στην ουσία προβλήματα. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι εξίσου σημαντικά και μπορώ να σας πω ότι ε, θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια ως προς ε, το κείμενο. Εάν θέλουμε μέχρι του χρόνου τον Ιούνιο να έχουμε ε, σωστά αποτελέσματα, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία refit φέτος. Πρέπει να, αξιολογηθεί, να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της διαβούλευσης φέτος, έτσι ώστε στην Γένοβα να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε μία πρόταση ε, πριν το Πάσχα του 2016. Αυτό είναι περίπου το χρονοδιάγραμμα. Και σε αυτό το χρονοδιάγραμμα θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και οι συγκητέ. από εσάς. Πρέπει λοιπόν να δοθεί η εντολή για τις ε, διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να καταφέρουμε να έχουμε όσο το δυνατόν συντομότερα, το πολύ στις αρχές του 2016, μια πολιτική συμφωνία. Αυτό είναι, προς, ε, αυτό είναι κάτι που θα είναι ωφέλιμο για όλους. Και πρέπει επίσης να δούμε και τα πλεονεκτήματα που μας δίνει η σαφήνεια. Όσο πιο σαφείς είμαστε, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει η δουλειά μας. Τώρα, ε, πνευματική ιδιοκτησία. Αναφερθήκατε σε αυτή, στο copyright και μας είπατε ότι πρέπει να δούμε το θέμα αυτό και από την σκοπιά του καταναλωτή και από, το, από τη σκοπιά της, ε, διαδικτυακής κοινότητας και όχι μόνο από τη σκοπιά του δημιουργού των ε, πνευματικών, ε, των έργων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, πρέπει να αναγνωριστεί και η ευθύνη των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, των εκδοτικών οίκων, και δεν, ε, δεν διατηρεί κάποιος ε, τα δικαιώματά του SAE, πρέπει να γίνεται συνέχεια αναθεώρηση. Εάν θέλουμε να υπάρχει ποικιλία στη μουσική, στο χώρο του βιβλίου, χρειάζεται να δημιουργηθεί και το κατάλληλο κλίμα. Χρειάζονται εκδοτικοί οίκοι, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, πλατφόρμες ε, ψηφιακές όπου θα προωθούν αυτήν την ε, ποικιλομορφία. Υπάρχουν επομένως τρεις πυλώνες και πρέπει και οι τρεις να δώσουν τη δική τους προστιθέμενη αξία. Τώρα αναφερθήκατε και στις εξαιρέσεις. Από τη μία υπάρχει το ζήτημα της φορητότητας ε, μετά της ε, διασυνοριακής ε, πρόσβασης και το γεωγραφικό ζήτημα εδώ χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ή να εξεταστεί έστω το θέμα και από την άλλη να γίνει και διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτά και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και στη χρήση του για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πρέπει να γίνει λοιπόν ο διαχωρισμός της πνευματικής ιδιοκτησίας ανάλογα με τον ε, τρόπο χρήσης της. Βέβαια, δεν είμαι σε θέση να λύσω εγώ τα δημοσιονομικά προβλήματα των κρατών ή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διασφάλιση της ε, ποιότητας, ιδιαίτερα στον ε, χώρο της εκπαίδευσης, είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ δεν ε, επιθυμώ μια επιδείνωση του επίπεδου. Θέλω το αντίθετο. Θέλω να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε, αν μπορούμε, τις Ηνωμένε Πολιτείε στην ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού και στην προσβασιμότητα, προσβασιμότητα σε αυτό. Σχετικά με το Euronews τώρα. Σίγουρα δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Και δεν μπορούμε να κόψουμε τον ομφάλιο λόρο με το ζόρι. Πρέπει να δώσουμε στο Euronews μία ευκαιρία. Συνομίλησα λοιπόν με τους τρεις κύριους ε, μετόχους, το ΡΑΙ και τους ε, Γάλλους Και βέβαια πρέπει να πω ότι ως Γερμανός λυπάμαι πολύ για το ότι η κρατική ραδιοτηλεόραση δεν επιθυμούσε καμία συμμετοχή. Προσπάθησα να συμπεριλάβω και την γερμανική ραδιοτηλεόραση. Δυστυχώς όμως παρά τις προσπάθειές μου δεν είδα καμία προθυμία. Όσον αφορά το Συμβούλιο για το πρόγραμμα. Αυτό πρέπει να είναι εξωτερικό και για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα. Ο προϋπολογισμός του Euronews επίσης πρέπει να εγκρίνεται από έτος σε έτος και όχι να γίνεται κάποιο καταποκοπήν ποσό για τα επόμενα χι χρόνια. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί σε ένα βαθμό η αντικειμενικότητα. Αυτό που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση είναι να δημιουργήσουμε ένα ε, φορέα της άποψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε ένα ανεξάρτητο Euronews όπου ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορεί να απολεμβάνει αντικειμενική ανταπόκριση και τηλεόραση. Και αυτό για να γίνει πιστεύω χρειάζεται, αναθε... χρειάζεται έγκριση κάθε χρόνο, έγκριση του προϋπολογισμού κάθε χρόνο. Αναφερθήκατε επίσης στο zero rating, στα χορηγούμενα δεδομένα της τηλεφωνίας. Το φθινόπωρο θα έχουμε νεότερα και τότε θα είμαι έτοιμος να τοποθετηθώ, να αναφερθώ σε αυτά που ήθελε ο νομοθέτης, σε αυτά που έγιναν δεκτά, σε αυτά που είναι εφαρμόσιμα και όχι. Αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο Σεπτέμβριο τον Οκτώβρη σε συνεργασία με την Προεδρία του Λουξεμβούργου. Επίσης αναφερθήκατε στο, στην προστασία των δικαιωμάτων της παροχής υπηρεσιών. Εδώ υπάρχουν διαφορέ στα κράτη-μέλη. Πιστεύω, για παράδειγμα, ότι στην Ισπανία βρίσκονται πολύ πιο μπροστά από ότι στη Γερμανία. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να νομοθετήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να δούμε όμως ε, τι θα γίνει. Όσον αφορά τώρα την ελευθερία στις ε, πανορομικές φωτογραφίες, να πω ότι οφείλουμε να σεβαστούμε την εθνική, τις εθνικές νομοθεσίες. Σίγουρα δεν είμαι υπέρ του περιορισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ προσωπικά ότι ό,τι μπορούμε να δούμε με, το, με τα μάτια μας, φύση, αστικό τοπίο, μνημεία, είτε αυτό είναι ένα δέντρο, είτε ένα δάσος, είτε ένας πύργος, είτε μια πλατεία. Αυτά λοιπόν, ό,τι μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να τα βλέπουμε και στο διαδίκτυο. Δεν πιστεύω πως χρειάζεται κάποιος περιορισμός. Παλαιότερα τραβούσαμε φωτογραφίες και τις είχαμε αυτές τις αναμνήσεις στο φιλμ. Τώρα το λογισμικό έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Και ας μην ξεχνάμε και τον ρόλο των κοινωνικών μέσων. Πιστεύω δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τη σημασία που έχουν πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Γαλλία και η Ιταλία είναι χώρες που έχουν πάρα πολύ πλούσια πολιτισμική κληρονομιά. Και δεν νομίζω ότι ζητά κανείς εκεί χρήματα για φωτογραφίες μνημείων που έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο. Η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από πολυμορφία. Πολυμορφία μέχρι και στην, ε, στο συγκεκριμένο αυτό θέμα, στις πανοραμικές φωτογραφίες. Δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από αυτά που συμβαίνουν σε κάθε κράτος μέλος, σίγουρα όχι από αυτά που γίνονται στη δική μου ε, χώρα, όμως δεν μπορούμε να ελέγξουμε με αυτόν τον τρόπο και να υποχρεώσουμε σε αποζημίωση. Πιστεύω πως δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθήσουμε καν. Νομίζω πως ε, με αυτό απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Παίρναμε τώρα στον επόμενο κύκλο ερωτήσεων. Σας παρακαλώ να τηρήσετε το όριο των δύο λεπτών ανά ευρωβουλευτής. Έξι μέλη έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριος Φίζας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Κυρία Κάμερπεργκ, αλλά και εσείς μιλήσατε για τα δικαιώματα που πρέπει να προστατεύονται και θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε τις προτάσεις της Επιτροπής ιδιαίτερα όσον αφορά την απαγόρευση κάποιων περιεχομένων αλλά και την προστασία των παιδιών, των ανηλίκων βάσει των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών. Και δεύτερη ε, σύντομη ερώτηση για τα αθλητικά. Τι λέτε για το δικαίωμα ενημέρωση σχετικά με αθλητικά αποτελέσματα σε σχέση με τα νόμιμα δικαιώματα των διοργανωτών των εκδηλώσεων αυτών, των διοργανώσεων αυτών. Μήπως υπάρχει ένα, μια σύγκρουση συμφερόντων εκεί, σας ευχαριστώ. Ήσασταν καταπληκτικός και εντός του χρόνου σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Λιμπάτσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον Επίτροπο και για την δέσμευση που αναλάβατε. Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ εγώ στον ψηφιακό κόσμο. Όσον αυτές οι δεξιότητες αυξάνονται, τόσο αυξάνεται και ο αποκλεισμός από τον κόσμο αυτό. Και φυσικά υπάρχει αποκλεισμός που οφείλεται στην γεωγραφική περιοχή, αλλά και σε κάποιες κατηγορίες πληθυσμών. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι δεν διαθέτουν αυτές τις δεξιότητες, που είναι αναλφάβητοι για τα ψηφιακά θέματα, είναι σήμερα θύματα αποκλεισμού. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να υιοθετήσουμε πρωτοβουλίες, για να εκπαιδεύσουμε, να καταρτήσουμε όλες αυτές τις κατηγορίες ε, προσώπων. Δεύτερη ερώτηση. Μήπως θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική η οποία να διευκολύνει την ε, κατάρτιση για πολύ στοχευμένες κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν παρακολουθούν το παραδοσιακό και επίσημο εκπαιδευτικό σχολικό σύστημα, οι οποίοι να μπορούν να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε κάτι για τις μικροπληρωμές. Αυτό το σύστημα των μικροπληρωμών θα μπορούσε ίσως να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ στο χρονοδιάγραμμα των προτάσεων της Επιτροπής όσον αφορά την οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα. Πότε μπορούμε να περιμένουμε την συγκεκριμένη πρόταση της Επιτροπής και δεύτερον, πώς βλέπετε να βελτιώνεται η προώθηση των ευρωπαϊκών ε, έργων Μιλήσατε για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Εγώ ήμουν ε, παρόν εκπρόσωπος της Επιτροπής μας στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Καρλό Βελεβάρη. Το ενδιαφέρον των νέων ήταν εντυπωσιακό. Είδα νέους οι οποίοι περίμεναν στην ουρά τέσσερις ολόκληρες ώρες για να αγοράσουν ένα εισιτήριο και να μπορέσουν να δουν αυτές τις ταινίες. Χρειάζεται λοιπόν βελτίωση της πρόσβασης σε αυτά τα κινηματογραφικά έργα για τους νέους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σρογιέσκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Έχω τρεις ερωτήσεις. το θέμα του περάσματος από το αναλογικό στο ψηφιακό σύστημα για το ραδιόφωνο. Πολλές χώρες έχουν ε, ήδη πάρει την απόφαση με πολύ διαφορετικό τρόπο. Μεγάλη αποτυχία στην Μεγάλη Βρετανία με αποτέλεσμα να υιοθετήσουν το σύστημα DAB και να το εγκαταλείψουν προτιμώντας το DAB2. Τι θέλω να πω, εθνικές λύσεις δεν είναι αποτελεσματικές ε, στον τομέα αυτό. Θα πρέπει σίγουρα να βρούμε ευρωπαϊκές λύσεις, ομοιογενείς λύσεις για όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν προτάσεις της Επιτροπής για τον τομέα αυτό, έτσι ώστε να μειωθεί και το κόστος και οι αποτυχίες. Δεύτερη ερώτηση, πώς συνεργάζεστε με τον Αρμόδιο Επίτροπο για τα οικονομικά θέματα. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι αρμόδιοι για τα οικονομικά θέματα δεν έρχονται εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού. Δέκα χρόνια έχουμε να δούμε τον αρμόδιο επίτροπο. Την ίδια ώρα οι επιτροπή αρμόδιοι για πολιτιστικά θέματα παίρνουν το λόγο στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και σαν αποτέλεσμα τα οικονομικά μέσα που διαθέτουμε, τα οποία δεν είναι πολύ σημαντικά, δεν είναι αρκετά. Αν συγκρίνει κανείς τη χρηματοδότηση για τον τομέα του πολιτισμού με αυτά που δαπανώνται για τη γεωργία διαπιστώνει ότι είναι πάρα πολύ ε, περιορισμένα. Όσον αφορά το διαδίκτυο, θα πρέπει να δούμε το διαδίκτυο σαν μία μεγάλη επιχείρηση. Οι στόχοι που θέτουμε εμείς δεν είναι καθόλου ρεαλιστικοί και σίγουρα θα πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος με τους φορείς του διαδικτύου. Ε, thank Σας ευχαριστώ, Επίτροπε, για τον διάλογο που συνεχίζουμε και έχουμε. Εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα για, την, για τα θέματα της κοινωνίας των πολιτών και για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη δουλειά σας. Διότι αν δεν διαβουλευτούμε επαρκώς την κοινωνία θα αισθάνεται εκείνη αποκλεισμένη από όλη τη δουλειά που κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανησυχώ ιδιαίτερα για θέματα που αφορούν στα παιδιά, στην ασφάλεια των παιδιών. και στον αντίκτυπο της ε, νομοθετικής ε, δουλειάς που κάνουμε επί των παιδιών και της ασφάλειάς τους ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά στο ίντερνετ. Επίσης θέματα θεμελιδών ε, δικαιωμάτων και ελευθερίας. Γνωρίζουμε για την ε, πρόσφατη απελευθέρωση του Ναμπίλ ε, Ρατζάντ και διάφορων bloggers που έχουν εχμαλωτιστεί και κρατούνται κτλ. Ε, πρέπει αυτά να λαμβάνουμε υπόψη μας όχι μόνο εντός των συνόρων μας αλλά και εκτός, παγκοσμίως δηλαδή. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, πτυχή της ε, ισότητας των φύλων σχετικά με το θέμα αυτό. Εγώ ήμουν από εκείνες που πήγαν στο ε, Διεθνές Σάμιτε για την πληροφορία, για την ενημέρωση στη Γενέβη και δεν μου άρεσε καθόλου ότι στις δηλώσεις υψηλών πολιτικών ηγετών και υπουργών δεν υπήρχε καμία γυναίκα ε, που να συμμετέχει στο μάνελ. Αυτό πρέπει να αλλάξει και πρέπει να είστε κι εσείς μέρος αυτής της διαδικασίας για σωστή εκπροσώπηση των γυναικών εντός της ψηφιακής οικονομίας καθότι <clears throat> εκπροσωπείτε και την κοινωνία και θέλω να μιλήσω και για τις ε, απομακρυσμένες περιοχές ε, της Υπέθρου και την κάλυψή τους στην ευρυζωνική. Εγώ εκπροσωπώ μια αγροτική κοινότητα της υπαίθρου. Έχουμε διάφορες μικροεπιχειρήσεις που δεν έχουν επαρκή διαδικτυακή κάλυψη και νομίζω ότι ε, εκεί θα άξιζε να δούμε και το έργο της Ίνκα που σε συνεργασία με την Ήψα ε, ε, προσπαθεί να αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους. Σας ευχαριστώ λέει η πρόεδρος, η κυρία Στροϊ... Ιώβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω Επίτροπε ότι περιγράψατε πληρέστατα το πρόγραμμά σας. Εγώ θα ήθελα να εστιαστώ κυρίως στην ταχύ ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες είναι εποφελείς, δίδουν ευκαιρίες για την βελτίωση της εκπαίδευσης για την καλύτερη πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά. Αλλά ενέχουν αυτά τους κινδύνους που ανέφερε και η κυρία Λιμπάτσκα και άλλοι συνάδελφοι και ε, θέτουν και το θέμα της ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών. Έχουμε τον κίνδυνο να προχωρήσουμε προς ε, μεγαλύτερες ανισότητες σε αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρούμε κατά νου το πρόβλημα αυτό και να προσπαθούμε πάντοτε να το αντιμετωπίζουμε εντός του πλαισίου των τηλεπικοινωνιών και, οπτικό, και διατάξεων επί του οπτικού ακουστικού. Θα πρέπει λοιπόν, πιστεύω, να βρούμε τρόπους εντός ε, της, του θεματολογίου 2020 να συμπεριλάβουμε περισσότερες ευάλωτες ομάδες, να τις εντάξουμε καλύτερα εντός των τεχνολογιών αυτών, εκεί όπου δηλαδή η αγορά η ίδια δεν επαρκεί, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχουμε στο επίπεδο των ε, ε, επενδύσεων δηλαδή. Για το Euronews και το Euronet συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι η αντικειμενική ενημέρωση επί των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Τα εθνικά μέσα ενημέρωσης τα δημόσια εθνικά μέσα ενημέρωσης δεν βλέπουν τις ευρωπαϊκές εξελίξεις ως υψηλής προτεραιότητας υλικό. Αυτό που θα ήθελα εγώ λοιπόν να δω θα ήταν μια πλατφόρμα αν θέλετε ενημέρωσης που να παρέχει αντικειμενική ενημέρωση, αντικειμενικές πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά ζητήματα αλλά θα πρέπει να ακολουθούμε κάποιε ελάχιστες αρχές. Θα ήθελα λοιπόν να δω το Euronews να μένει εντός συγκεκριμένων αρχών και αξιών και κανόνων. Όπως βλέπετε επίτροπε οι συνάδελφοι παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον και θέτουν πολλά ερωτήματα. Εσείς διακρίνατε ε, το δικαίωμα ευρεστεχνίας αν θέλετε από το πνευματικό δικαίωμα. Δηλαδή έχουμε εδώ διαστάσεις και οικονομικές και πνευματικές ιδιοκτησίες και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και η έρευνα που θα γίνει σχετικά με την ε, σωστή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων, αν θέλετε, των χρηστών και των δικαιωμάτων των δημιουργών. Αυτών δηλαδή που ζουν από αυτό το επάγγελμα, από αυτήν την επαγγελματική δραστηριότητα. Και ε, εξ όσων προκύπτουν και ίσως και στο πλαίσιο της ε, ψηφιακής πολιτικής της Κομισιόν υπάρχει μια υπογράμμιση περισσότερο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρά της ηλεκτρονικής κοινωνίας των πολιτών, για να την πούμε έτσι, της, εν πάση περιπτώσει της e-citizenship, του τρόπου με τον οποίο μπορούν να εκφράζονται ψηφιακά, δηλαδή ενδιαφερόμενοι φορείς. Τρίτον, για την VNS, την οδηγία, την επανεξέταση, εμείς ε, θεωρώ και επιτρέψτε μου να πω ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο εντός της χρησιμοποίηση αυτής της μεγάλης τράπεζας δεδομένων που είναι το παρατηρητήριο οπτικοακουστικού υλικού του Στρασβούργου που ονομάζεται Μαρβί, το γνωρίζετε δίχως άλλο επίτροπε και εκεί σημειώνεται ότι υπάρχει κίνδυνος μείωσης χρηματοδότησης και είναι η μοναδική πηγή ενημέρωση που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις εκπομπές οπτικοακουστικού υλικού. Και ε, κλείνω λέγοντας ότι και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθεί κανένας διαφάνεια στο Euronews αλλά δεν πρέπει μαζί με τα χαλασμένα φρούτα να πετάξουμε και τα φρέσκα όπως θα λέγει κανείς. Ε, υπάρχει όμως ένας κίνδυνος να υπάρξει μια ανισορροπία και έχουμε και κάποιες φορείς που δεν δρούν πάντα με απολύτως διαφανή, διαφανείς προθέσεις. Χρειάζεται λοιπόν επαλήθευση, χρειάζεται έλεγχος, αλλά χρειάζεται και έλεγχος επί των λοιπόν broadcaster όλων των χωρών για να έχουμε σωστή ισορροπία. Παρακαλώ. Καταλαβαίνω πολύ καλά τις ανησυχίες σας, τις ακούω και πραγματικά έχω εμπιστοσύνη σε αυτά που γίνονται όσον αφορά τις προσδοκίες των Ευρωπαίων είμαι σίγουρος ότι οι εξελίξεις θα ακολουθήσουν αυτές τις προσδοκίες και φυσικά εμείς παρακολουθούμε και αξιολογούμε τα προγράμματα ακούμε τις διαμαρτυρίες και τα παράπονα και τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Όλοι όσοι μίλησαν έδειξαν ότι συζητάμε θέματα ρυθμιστικά, κανονιστικά, που φυσικά είναι πολύ ενδιαφέροντα από άποψη τεχνολογική, αλλά και κοινωνική, που είναι στην επικαιρότητα, που καλύπτουν πολλούς τομείς και που περιέχουν και πολλούς κινδύνους. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε ευρωπαϊκά. Αυτή είναι η σωστή επιλογή. Και πρέπει να δούμε στα πλαίσια της επικουρικότητας τι είναι καλύτερο να κάνουμε. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό copyright, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό δικαίωμα προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού και δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή αξιολόγηση κανένας ευρωπαϊκός ορισμός όσον αφορά την ουδετερότητα των δικτύων. Μπορούμε να λέμε λοιπόν ό,τι θέλουμε, αλλά εμείς σαν Ευρωπαίοι μπορούμε να κάνουμε πολλά εάν λάβουμε υπόψη μας την επικουρικότητα. Η ψηφιακή επανάσταση θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να είμαστε προσεκτικοί και να παρακολουθούμε αυτά που συμβαίνουν. Προστασία των νέων Καταλαβαίνω πολύ καλά την ανησυχία σας και φυσικά και υπάρχουν σήμερα διαφορετικά όρια προστασίας για τους νέους για τους ανήλικους. Εγώ καταλαβαίνω ότι η τεχνολογική εξέλιξη στον ψηφιακό κόσμο δημιουργεί προγράμματα τα οποία εκπέμπονται χωρίς κανένα φραγμό. Έχει νόημα λοιπόν σήμερα να μιλάμε για προστασία των νέων. Είναι πολύ σημαντική η ιδέα ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά γιατί αυτό είναι τμήμα της αποστολής μας για την εκπαίδευση των νέων. Και φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητούν και οι ε, οικογένειες αλλά και οι κοινωνίες. Είναι ε, ε, ο ρόλος του νομοθέτη. Το θέμα όμως είναι ότι τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης ε, βεβαίω ε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουν ένα ρόλο προστασίας των ε, νέων. όταν όμως δεν πρόκειται για επιχειρήσεις, για κανάλια, για τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά για πλατφόρμες, πώς μπορούμε να μιλήσουμε για αυτήν την υποχρέωση. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να γίνει ανάλυση αυτών των ε, δεδομένων της πλατφόρμας, να ξέρουμε πολύ συγκεκριμένα πώς γίνονται οι αναμεταδόσεις και άκουσα που είπατε ότι εδώ υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα και αντικρώμενα συμφέροντα. Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε παραδείγματος χάρη το θέμα του, ε, ε, των ποδοσφαιριστών που φεύγουν από τη Βραζιλία και πάνε στη Βαρκελώνα, στο Μόναχο, στο Μάντσεστερ. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί κερδίζουν περισσότερα χρήματα. Τα χρήματα αυτά βεβαίως όταν μιλάμε για τηλεοπτικές εκπομπές, από πού προέρχονται, από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο, από τον Ευρωπαίο τηλεθεατή, ο οποίος πληρώνει την συνδρομή του, πληρώνει φόρους και βεβαίως και από την διαφήμιση. Το θέμα είναι ότι η διαφήμιση οδηγεί στο να αγοράσουμε κάποια προϊόντα, Adidas, Mercedes, Peugeot, Nike. κρασί γαλλικό ή σαμπάνια, γκούτσι ή πράντα κτλ. κτλ. Πρόκειται λοιπόν για κάποια συμφέροντα τα οποία εμείς πρέπει να εντοπίσουμε και να προχωρήσουμε στην ρύθμιση αυτών των τομέων. Δεν μιλάμε για τον αθλητισμό και για τα ε, κέρδη. Πρέπει να δούμε όλη την αλυσίδα πρόθεση αυτών των προϊόντων στον αγορά. Φυσικά είναι πολύ σημαντική η Real, η Μπάρσα. Και φυσικά είναι πολύ σημαντική και η γεωγραφική, αν θέλετε, ο γεωγραφικό εντοπισμό αυτών των συμφερόντων. Αυτό που θέλουμε δεν είναι απλώς μόνο οι επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές να προστατεύονται και να ρυθμίζονται ε, στον χώρο που δραστηριοποιούνται. Αλλά το ίδιο και για το handball, το ίδιο και για άλλα αθλήματα τα οποία είναι λιγότερο εμπορικά. Δεν υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μία αγορά. Αν θέλει παραδείγματος χάρη κάποιος να προστατεύσει τον αυστριακό κινηματογράφο χρειάζεται για την Βιέννη, για την αγορά όλη της Αυστρίας, για τη γερμανική αγορά, για την ελβετική γερμανόφορη αγορά, έτσι ώστε ένα, μια ταινία από την Αυστρία να μπορεί να, κινητο, να κινητοποιήσει και τηλεθεατές και ακροατήριο από άλλες χώρες. Γι' αυτό και μιλάμε εδώ για τις εξαιρέσεις όσον αφορά την ε, πολύ συγκεκριμένη αφενός γεωγραφική ε, διάδοση γιατί ξέρετε ότι αλλιώς το Hollywood θα κατακλείσει όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε κίνητρα προώθηση στον κινηματογράφο τον ευρωπαϊκό και αυτό θα προγίνει σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν θέλουμε να υπάρξει περαιτέρω κατηγοριοποίηση και αποκλεισμό κάποιων συγκεκριμένων κατηγοριών Ευρωπαίων πολιτών χρειαζόμαστε κατάρτιση, χρειαζόμαστε υποστήριξη έτσι ώστε όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση αλλά και δεξιότητες σε αυτό το νέο ψηφιακό κόσμο. Και φυσικά και χρειάζεται ε, κατάρτιση, χρειάζονται παραδείγματος χάρη συγκεκριμένη, αν θέλετε, κατάρτιση να επιτρέπει σε αυτούς οι οποίοι είναι εκτός του παραδοσιακού σχολικού εκπαιδευτικού συστήματος και οι οποίοι όμως έχουν πρόσβαση μέσω των smartphone, μέσω των ε, ε διαφόρων άλλων ηλεκτρονικών μέσων σε υλικό το οποίο μπορεί να είναι και εκπαιδευτικό υλικό. Γνωρίζουμε όλοι ότι σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Το θέμα είναι όμως να μην χάσουν οι ευρωπαϊκοί φορείς, η Ευρώπη με ευρωπαϊκούς φορείς θα πρέπει να αποκτήσουν και την δυνατότητα να προστατεύσουν την ταυτότητά τους. Έχουμε επαφή με πολύ σημαντικούς φορείς ε, του τομέα. Εγώ πήγα σε τέσσερις διαφορετικές εκθέσεις φέτος που εκπροσωπούνται όλοι οι πολύ συγκεκριμένοι φορείς και επιχειρήσεις αυτού του κόσμου και φυσικά μας ενδιαφέρουν τα connecting cars, τα συνδεδεμένα δηλαδή αυτοκίνητα, όλος ο κόσμος της αυτοματοποίησης Και συχνά οι εθνικές πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό γίνονται ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες αν στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες. Και αυτό βεβαίως το είδαμε στην Πορτογαλία, στη Σλοβακία, στη Γερμανία. Πρέπει να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία να βοηθήσουν στην πρόθεση αυτών των προϊόντων. Βεβαίως και εγώ είμαι σε στενή επαφή με τους φορείς στον τομέα του πολιτισμού και θέλω να ενισχύσω τον τομέα αυτό. Δεν υπάρχει εδώ πόλεμος με τους αρμόδιους επιτρόπους για τα οικονομικά θέματα. Πρόκειται για την κληρονομιά μας, την οποία θα πρέπει να στηρίξουμε. Και όσον αφορά αυτό που είπατε για τη γεωργία, δεν μπορεί εδώ να υπάρξει αντιπαράθεση μεταξύ της υπαίθρου του αγροτικού κόσμου και του πολιτισμού. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να το δούμε σαν σύγκρουση συμφερόντων. Προς συμφέρον της ε, ανάπτυξης και του αγροτικού κόσμου θα πρέπει να στηρίξουμε τον πολιτισμό. Είναι επίσης πάρα πολύ ε, σημαντικό να δούμε ότι οι τομείς αυτή των τεχνολογιών είναι τομείς που γίνονται διακρίσεις όσον αφορά το φύλλο. Εκπροσωπούνται σε όλους αυτούς τους τομείς, τους μηχανικούς αλλά και στον τομέα της πληροφορικής πολύ περισσότεροι άντρες από γυναίκες. Χρειάζεται όμως δημιουργικότητα, χρειάζονται γυναίκες, χρειάζονται περισσότερες γυναίκες σε όλους αυτούς τους τομείς επιγόντως. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες σας και καλή τύχη. Thank you so much, uh, For... Ευχαριστούμε, πίτροπε για την γενεοδορία σας και για όλο το χρόνο αυτό που μας αφιερώσατε. Εμείς θα παραμείνουμε σε τακτική, συνεχή επαφή μαζί σας και θα παρακολουθούμε τις υπόλοιπες συναντήσεις στα πλαίσια αυτής της ατζέντα. And now the, the last effort. <laughs> Sorry, because we have uh, two important people. Τώρα έχουμε ακόμα δύο γνωμοδοτήσεις, λέει η Πρόεδρος. Και για να είμαστε εντός των χρονικών ορίων, θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο που είναι η εισηγητής για τα θέματα ριζιστο... ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγηση Ευρωπαίων πολιτών από κινήματα φονταμενταλισμού στον κύριο Τζαμπάσκι. Ε, σημαντική έκθεση που θα υποβληθεί και στην ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Αύριο έχουν προγραμματιστεί οι τροπολογίες. Δεν γινόταν διαφορετικά εν ώψη των θερινών διακοπών. Και θα έχουμε ψηφοφορία στις 15 Σεπτεμβρίου στην Κούλτ και αμέσως μετά στην ε, Λίμπε. Α, στις 12 Οκτωβρίου στη Λίμπε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς να ευχαριστήσω για την δυνατότητα αυτή που έχω σήμερα να σας παρουσιάσω αυτήν την, ε, αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης της ρίζος παστικοποίησης και των κινημάτων φονταμενταλισμού είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις ε, χώρες μέλη και πρέπει να το συζητούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. Η στρατολόγηση πολιτών προκειμένου να πολεμήσουν κατά των πιο θεμελιωδών αξιών και αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ταχύτατα. Και ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης. Ε, τον Μάρτιο φέτος υπεγράφει η διακήρυξη του Παρισίου η οποία προβλέπει μια ενισχυμένη συνεργασία στο επίπεδο των θεμελιωδών αξιών με τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαφορετική προστασία στη διαφορετικότητα Πρέπει εκτός από την επισήμανση του προβλήματος, να καταπολεμήσουμε τα αίτια του. Με την ψηφιακή τεχνολογία σήμερα η διάχυση οποιοδήποτε μηνύματος είναι, έχει καταστεί πανεύκολη. Αυτό είναι ακόμα πιο προβληματικό όταν αυτή η διάχυση μπορεί να μεταφέρει μηνύματα βίας και εξτρεμισμού. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε όλα τα επίπεδα που μπορούν να εκπαιδεύσουν καλύτερα και να αποτρέψουν το οικογενειακό, το σχολικό και υπάρχουν ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες μεταξύ του πληθυσμού προς τέτοιου είδους μενήματα που είναι οι νέοι. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε μέτρα κατά της περιθωριοποίησης σε εθνικό βεβαίως επίπεδο αλλά η Κομισιόν θα πρέπει να ηγείται των προσπαθειών ε, σχετικά με τη χρησιμοποίηση ε, μέσων χρηματοδότησης εκτάκτου ανάγκης για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης. Στα πλαίσια της προετοιμασίας της γνωμοδοτήσεώς μου βλέπουμε τις ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν και θα ήθελα να προτείνω επίσης την προσθήκη μιας τροπολογίας στην γνωμοδότησή μου δηλαδή σχετικά με τα προγράμματα σπουδών των σχολικών μας ε, ιδρυμάτων, γιατί σε μερικές περιπτώσεις ιδιωτικών μουσουλμανικών σχολείων ενσωματώνονται στα προγράμματα σπουδών εξτρεμιστικά κείμενα και βιβλία τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακριβώς σε τέτοια φαινόμενα ριζοσπαστισμού. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω, μιλώντας κυρίως για την έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ σχετικά με το θέμα αυτό, για την χρησιμοποίηση της εκπαίδευσης ως μέσο εξτρεμισμού και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ και στις ε, πολύ δυσάρεστες αρνητικές συνθήκες που ισχύουν στις φυλακές και τα κέντρα κράτησης. Και εκεί είναι ένας χώρος με τον οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε. νομίζω ότι με το σύνολο των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί θα μπορέσουμε να υποβάλουμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ μία γνωμοδότηση με συγκεκριμένες απτές προτάσεις για τα θέματα τουλάχιστον πολιτισμού και εκπαίδευσης. Η προθεσμία είναι στις 15 Ιουλίου το μεσημέρι. Το μεσημέρι και ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι οι σκιώδεις θα έχουν ε, μέχρι τότε το χρόνο να συζητήσουν διεξοδικά για συμβαστικές προτάσεις τροπολογιών. Εγώ θα παρουσιάσω τις δικές μου την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου η ταχύτητα βεβαίω εξηγείται από το γεγονό ότι θα πρέπει εγκαίρω να δώσουμε, να διαβιβάσουμε αυτή τη γνωμοδότηση στην αρμόδια επιτροπή για να προλάβει και εκείνη με τη σειρά τη να κάνει τη δουλειά τη εγκαίρω. Και επαναλαμβάνω, ότι πρόκειται για μια επίγουσα ανάγκη πρώτης κατηγορίας θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δουλέψουμε και μάλιστα επί ενός προτύπου ανταλλαγής βελτίστων πρακτικών σχετικά με τα μέτρα που μπορούμε να αναλάβουμε στις χώρες μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και θα έχουμε και ακρόαση επί του θέματος αυτού. Η κυρία Σβέρ καταρχάς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Οφείλω να ομολογήσω πως χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι η Επιτροπή Πολιτισμού είχε την ευκαιρία να συντάξει μια γνωμοδότηση στην έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Εκ πρώτης όψεως το θέμα αυτό φαίνεται πως αφορά την ασφάλεια και μόνο. Όμως, εάν πραγματικά θέλουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα, πρέπει να το αναλύσουμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες και εδώ έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουμε. Πιστεύω ότι ο κύριος Τζαμπάτσκι ετοίμασε μια εξαιρετική γνωμοδότηση. Εμείς θα την εμπλουτίσουμε με τις ε, τροπολογίες μας και ελπίζω μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουμε ένα καλό κείμενο. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Η Ευρώπη έχει πολλά θέματα τα οποία οφείλει να επιλύσει. Τα θέματα αυτά δεν θα είχαν γίνει προβλήματα μεγάλα εάν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν εκείνοι που συμμετείχαν σε τρομοκρατικές ενέργειες και εντός και εκτός της επικράτειας της Ένωσης. Και ο ρόλος μας είναι να αποτρέψουμε ακριβώς αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση, να αποτρέψουμε τη στρατολόγηση. Έχουμε ανάγκη από ένα σύστημα το οποίο θα αποτρέπει τη στρατολόγηση. Φυσικά μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα από διάφορες οπτικές γωνίες, από την δικαστική άποψη, όπου παρατηρούμε πως πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος ορισμένων οργανισμών, Europol, Eurojust για παράδειγμα, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα σύστημα ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών. Έχουμε ήδη συζητήσει διάφορου τρόπου με του οποίου μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Και ορισμένα κράτη-μέλη επιβάλλουν ήδη κυρώσει στου ε, λεγόμενους ξένου μαχητέ. Και με τον τρόπο αυτό θα αποτρέψουμε άλλους πολίτες της Ένωσης από το να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και να πολεμούν στο πλευρό αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος όμως καταπολέμησης του προβλήματος αυτού είναι η παιδεία, η εκπαίδευση, τα σχολεία, αλλά όχι μόνο αυτά. Πρέπει να συμπεριληφθούν πολλά στοιχεία δημοκρατίας την διδακτέα ύλη των ε, σχολείων. Πρέπει να εξεταστούν τα συμβάντα του παρελθόντος για να δούμε και να διδαχθούν οι μαθητές το τι πρέπει να αποφύγουμε. Έτσι θα δημιουργηθεί συνείδηση για να αποφευθεί η ριζοσπαστικοποίηση. Όμω, όπω σα είπα, τα σχολεία δεν είναι οι μόνοι φορεί που μπορούν να συνεισφέρουν και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχουν σημαντική συμβολή. Τα μέσα ενημέρωσης επίσης έχουν σημαντικό ρόλο. Επίσης οι διάφοροι φορείς εμπειρογνωμοσύνης έχουν να συνεισφέρουν. Το φαινόμενο των ξένων μαχητών είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και για να αποφύγουμε και να αποτρέψουμε τη ριζοσπαστικοποίηση χρειάζεται ολιστική προσέγγιση. Χρειάζεται εκπαίδευση, σωστή εκπαίδευση και ακριβώς στο ρόλο της εκπαίδευσης εμείς έχουμε ένα λόγο. Έχουμε ακόμα μόνο 10 λεπτά διερμηνίας λέει η Πρόεδρος. Όχι, Τη διορθώνει κάποιος. Δεν έχουμε μόνο 10 λεπτά διερμηνίας, λέει τώρα η Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης διότι η Επιτροπή Πολιτισμού θα πρέπει να έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός έχουν πολύ σημαντική θέση και στην αποτροπή της ε, ε, παστικοποίησης όπως και της στρατολόγησης ε, Ευρωπαίων πολιτών προς ή από εξτρεμιστικές ομάδες. Νομίζω ότι εδώ απαιτείται μια προσέγγιση πολυεπίπεδη, καινοτόμα και τακτική, μόνιμη. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι η Επιτροπή μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη ακριβώς για την παρακολούθηση αυτών των τριών επιπέδων και θα πρέπει να έχουμε συνεχή συνεργασία μεταξύ διαφόρων ε, φορέων που συνεισφέρουν στην παρακολούθηση των ατόμων της οικογένειας όπως υπογράμμισαν και οι συνάδελφοι των σχολικών ε, ιδρυμάτων και των άλλων φορέων και οργανισμών έτσι ώστε να καταπολεμούνται τα αίτια στην ουσία των φαινομένων αυτών που είναι η περιθωριοποίηση, η φτώχεια, η πρώιμη εγκατάλεψη των σχολικών σπουδών. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει λοιπόν να εστιαστεί τα προγράμματα του σε δραστηριότητες που αφορούν διαπολιτισμικές αξίες. Αυτό το σλόγγαν, αυτό το μήνυμα θα πρέπει να επανέλθει σε κεντρικό σημείο στην προσοχή της πολιτικής μας ε, με ισχυρή εστίαση στην ενσωμάτωση χρησιμοποιώντας μάλιστα ακριβώς τις ψηφιακές ε, τεχνολογίες και τα social media ώστε να διαδίδεται στα σχολεία η υπεύθυνη χρησιμοποίηση των κοινωνικών media η υπεύθυνη χρησιμοποίηση της γλώσσας και των μηνυμάτων που περνούμε ώστε να μην είναι βία και να μην είναι υπέρ του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό πρέπει να γίνει η πρακτική σε όλα τα κρατη διότι αλλιώς θα συνεχιστεί αυτή η περιθωριοποίηση, θα έλεγα η γκαιτοποίηση που βλέπουμε σε πάρα πολλές χώρες. και αλλιώς θα έχουμε πολύ αυξημένο κίνδυνο, ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Θα πρέπει επίσης να εστιαστούμε στην ε, σωστή διδαχή των διαφόρων ε, ε, θρησκευτικών αν θέλετε, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο των οποίων πολύ συχνά βλέπουμε ότι παρισφρίουν εξτρεμιστικά μηνύματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να προσέχει όλα αυτά τα συστατικά θα πρέπει να είναι ένας καρπός μία σωστή ακαδημαϊκής και παιδαγωγικής προσέγγισης που να διέπεται και να ηγείται από εμπειρογνώμονες, από ειδικού. προκειμένου να αποφύγουμε και το φαινόμενο της ε, προσέλκυσης νέων προς ε, ριζοσπαστικά κινήματα και προκειμένου αυτοί που έχουν ήδη προσελκυστεί από τέτοια κινήματα να μπορέσουν να επανέλθουν αν θέλετε στην κοινωνία. Αυτό ιδιαίτερα για άτομα που προέρχονται από συγκεκριμένες οικογενειακές καταστάσεις, όταν δηλαδή αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα αποκλεισμού, τη διαβίου μάθηση που θα πρέπει να είναι μια συνεχής προσπάθεια και διαδικασία, όλα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλα κίνητρα που θα πρέπει να δίδονται στα άτομα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο για να μπορούν να αισθάνονται όλοι οι πολίτες μέρος, τμήμα της κοινωνίας και της ανάπτυξής της. Εγώ πάντως είμαι πολύ ικανοποιημένη που η Επιτροπή μας έχει την ευκαιρία να δουλέψει σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο μας θα πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά αυτή, το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και θα πρέπει πάνω απ' όλα να το παρακολουθήσουν τα κράτη-μέλη. Γιατί δυστυχώς όταν μιλούμε για τέτοια θέματα μιλούμε για τρομοκράτες, φανατικούς, αλλά δεν μιλούμε για το ίδιο το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης. Και για να το κατανοήσουμε πρέπει να κατανοήσουμε τις αιτίες του και να δώσουμε λύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Τόμ. Thank mm, ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ομολογώ πως ε, δεν είναι ένα θέμα που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Δυστυχώς. Ο συνάδελφος όμως έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Προσωπικά θεωρώ πως υπάρχει κάποιος ε, κίνδυνος όταν προσπαθούμε με τόση ζέση να καταπολεμήσουμε κάτι, ενδεχομένως ε, κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Κάνουμε πιο ορατό αυτόν τον κίνδυνο. Χρειάζεται λοιπόν ε, προσοχή και λεπτότητα στην διαχείριση του προβλήματος αυτού και από ό,τι φάνηκε από τις διαβολεύσεις στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, χρειάζεται ένα κοινωνιολογικό προφίλ αυτών των ανθρώπων. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, δεν ξέρουμε ε, αν ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, αν είναι περιοθωριοποιημένοι. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη κατανόηση του ιστορικού αυτών των ατόμων και σίγουρα Πιστεύω πως χρειάζεται να στηρίξουμε προγράμματα τα οποία θα προωθούν την ανεκτικότητα και χρειάζεται να ανταλλάξουμε βέλτιστες προοπτικές. Ιδιαίτερα για να αποτραπεί ο κοινωνικός αποκλεισμός των μεταναστών, των προσφύγων που έχουν έρθει πρόσφατα. Η δική μου εμπειρία από τη χώρα μου, την Εστονία, είναι ότι οι πολίτες δεν είναι τόσο ε, έτοιμοι να καλωσορίσουν κάτι το διαφορετικό. Χρειάζεται λοιπόν να προωθηθεί αμοιβαία συνεργασία, αμοιβαία κατανόηση και η συνεργασία των Ευρωπαίων ηγετών. Και σίγουρα πρέπει να αποφύγουμε να εισέλθουμε σε έναν προπαγανδιστικό πόλεμο. Χρειάζεται να συμφωνήσουμε για έναν κοινό κώδικα δεοντολογίας του τύπου και ως ε, δημοσιογράφος η ίδια πρέπει να σας πω ότι ο κώδικας δεοντολογίας έχει λόγο ύπαρξης και έχει αποτελέσματα. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργηθεί νομοθεσία, να δημιουργηθούν ποινές ε, για την ε, ρητορική μίσους και να γίνουν σαφείς ορισμοί. Προσωπικά θεωρώ πως πολλές φορές ε, η ελευθερία της έκφρασης είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται καταχρηστικά από κάποιες ομάδες και ίσως μου διαφεύγει ε, ο συνδετικός κρίκος με το τι γίνεται στα σχολεία, με τη βία στα σχολεία, με διάφορες ε, εγκληματικές ενέργειες που γίνονται εκεί, όμως μην στεκόμαστε μόνο στις άσχημες εμπειρίες. Έχουμε και ε, πολύ θετικές εμπειρίες, τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εξίσου. Σας ευχαριστώ. Εύανες παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο εισηγητής έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Όπως είπε η έκθεση για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είναι συνοπτικότατη και είχε και τους περιορισμούς που είχε και υπό το πρίσμα αυτή θα πρέπει να την βλέπουμε. Εγώ είμαι από την Ουαλία που είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, το συζητούμε αυτό πολύ στην Ουαλία σχετικά με τους νεαρούς ανθρώπους και ιδιαίτερα τις νεαρές γυναίκες που φεύγουν προς μέρη όπως η Συρία. Πάντως αντλώντας από την δική μου τουλάχιστον προσωπική εμπειρία υπάρχει, δεν έχει υπάρξει μάλλον μια συνεπής διαφοροποίηση μεταξύ της πρόληψης στην προσέλκυση σε τέτοιες οργανώσεις και στην αποτροπή εγκληματικών πράξεων, που είναι δύο διαδοχικά επίπεδα αν θέλετε. θα έλεγα λοιπόν ότι επί τη βάση αυτών που ήδη σημειώνει η γνωμοδότηση, στο πρώτο της τμήμα θα πρέπει να προσθέσουμε ότι δεν είναι απλώς η διακήρυξη των Παρισίων δηλαδή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει όμως να συμπληρώσουμε ότι μαζί με την προστασία της ασφάλειας και των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προασπίζει και την βασική αξιοπρέπεια και τη θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Αυτό που καθιστά πολύ συχνά κοινότητες ευάλωτες είναι ακριβώς τα φαινόμενα αποκλεισμού και περιθωριοποίησης. Ο ρόλος της εκπαίδευσης όπως λέει και ο εισηγητής είναι κρίσιμος εδώ. Γιατί εκεί ακριβώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις βασικές μας αξίες, τις βασικές μας αρχές και να, αν θέλετε, να αμφισβητήσουμε ή να βρούμε έναν τρόπο να συζητήσουμε ανοιχτά, εν πάση περιπτώσει, τα αίτια αυτής της ε, περιθωριοποίησης και κυρίως της ριζοσπαστικοποίησης και να αναγνωρίσουμε ότι πολλά άτομα μπορούν να προσελκυθούν προς τέτοιες τάσεις εξτρεμιστικές αλλά υπάρχουν διάφορες λύσεις και διάφοροι τρόποι να το συζητήσει κανείς και να το αντιμετωπίσει κανείς. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη με, κά... με κάποιες προσπάθειες και προγράμματα στρατηγικής exit, exit strategy δηλαδή, από τέτοιες οργανώσεις, δηλαδή από προσέλκυση των ανθρώπων από τέτοιες εξτρεμιστικές οργανώσεις. Και αυτό μπορούμε μόνο να το κάνουμε με, με ανθρώπους που θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι αλλά προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως, αν ποτέ θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως αυτά τα φαινόμενα, θα πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνουν. Και άρα δεν μπορούμε να ξεχνούμε τα όσα συμβαίνουν μεταξύ άλλων στη Συρία, τη βία του πολέμου, τις μεταναστευτικές ροές, τους πρόσφυγες, Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το πλαίσιο στο οποίο γεννώνται αυτές οι τάσεις δηλαδή. Αυτό εννοώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ward και μετά η κυρία Ζοϊντρόβα. Πρόεδρε, υπάρχουν πολλά κοινά σημεία επαφής ε, με τη δουλειά που κάνω εγώ, που προετοιμάζω εγώ για την διαπολιτιστική εκπαίδευση και με βοηθούν και αυτά που αναφέρετε και εσείς. Αναφερθήκατε σε κάποιους οδηγούς σπουδών, σχολικά βιβλία και θρησκευτικά προγράμματα εκμάθησης. Υπάρχει ένα κολέγιο στα βόρεια ανατολικά της Αγγλίας που ακολουθεί αν θέλετε μία τάση ε, αυτών που αποκαλούνται creationists. Αυτό με ανησυχεί εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι πρέπει να αναφέρουμε και άλλες θρησκείες εκτός από το Ισλάμ και τη μουσουλμανική θρησκεία όταν αναφερόμαστε σε ριζοσπαστικά και εξτερμιστικά κινήματα. Υπάρχουν και χριστιανικές θρησκευτικές οργανώσεις που δρούν προς την κατεύθυνση αυτή. Και μόλις τώρα έλεγχα λίγο στον υπολογιστή μου, ε, έβρισκα πληροφορίες σχετικά με την ομάδα αυτή, την τάση αυτή. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικά αυτά που διδάσκουν. Και οι, οι σπουδαστές, ας πούμε, αυτής της σχολής αποφυτούν με ιδέες εξαιρετικά στρεβλωμένες σχετικά με την πραγματικότητα και την προέλευση του κόσμου. Πρέπει να έχουμε μια ισόρροπη άποψη πιστεύω συνολικά για τα πράγματα. Σας ευχαριστώ ο κύριος Μαραγάλ. Πρόεδρε ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος έκανα λάθος στη σειρά. Δεν πειράζει, μιλήστε εσείς πρώτα κύριε Μαραγάλ. Εγώ συμφωνώντας απολύτως με τις παρεμβάσεις των συναδέλφων σχετικά με το ρόλο των ε, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των διδασκάλων, των βιβλίων του υλικού, διερωτώ με μήπως τονίζουμε υπερβολικά την πτυχή της απρολήψεως. Αντί να έχουμε αν θέλετε μια ματιά προοπτικής. Γιατί όσο καλύτερα κάνουν τη δουλειά τους τα σχολεία, τόσο περισσότερο θα μπορούσαμε, για να το πω έτσι, να πεθάνουμε από υπερβολική επιτυχία. Δηλαδή αυτό που λέμε ολιστική προσέγγιση τι σημαίνει. Σημαίνει δουλειά. Σημαίνει κοινωνική ένταξη, πολιτιστική, καλλιτεχνική, οικονομική ένταξη. Και φτάνει ένα σημείο στη ζωή, στα 14-16 χρόνια της ηλικίας, όπου η προσπάθεια που γίνεται στο σχολείο, που ήδη γίνεται αλλά πρέπει να βελτιωθεί, με εκπαιδευτικά προγράμματα των τοπικών και περιφερειακών αρχών που πρέπει να τις, ε, προφανώς να τις βοηθήσουμε με απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα όπου αυτή η σχολική εκπαίδευση μπορεί να καταλήξει σε μια αντίφαση γιατί τελικά όλα αυτά που λέμε στα παιδιά τους τα αρνούμεθα αμέσως μετά. Ένταξη, επιτυχία, όλα αυτά. Μετά τους λέμε ξέρετε κάτι, όλα αυτά it's not true λέει ο μιλητής. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αποκλειστική αλήθεια και, μία αποκλειστική, και καμία αποκλειστική ευθύνα Υπάρχουν κάποια πρότυπα οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Γνωρίζω τώρα ότι αναφέρομαι σε πράγματα που ξεπερνούν κατά πολύ τα πλαίσια και τα αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Αλλά ακριβώς ο ρόλος μας πιστεύω ότι είναι να, να θέτουμε τέτοια ζητήματα και προς άλλες επιτροπές. Ιδάλλως, παγιδεύουμε τον εαυτό μας σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Ζευντρόβα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Στην ουσία αυτό που ζητούμε είναι να δημιουργήσουμε μέσα που θα αποδειχθούν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, η οποία πρεσβεύει κάποιες απόψεις οι οποίες απορρέουν από την πεποίθηση ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Δείχνει λοιπόν μια δυσλειτουργία της κοινωνίας μας. Όταν υπάρχουν ε, οικογενειακά περιβάλλοντα που είναι άσχημα, όταν οι οικογένειες δεν είναι μονάδες μιας ευρύτερη κοινωνίας, όταν Υπάρχουν οικογένειες που εξαρτώνται από την κοινωνική πρόνοια. Αυτά είναι λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Ε, η εκπαίδευση, λέτε, θεωρείται ε, το μέσο καταπολέμησης της ε, ριζοσπαστικοποίησης. Ας δούμε λοιπόν τι μέσα διαθέτει η εκπαίδευση. Συνήθως το προφίλ ενός ριζοσπαστικοποιημένου ατόμου ε, έχει καλό μορφωτικό ε, επίπεδο. Όμως εκείνη που προσιλητίζει όχι. Χαρακτηρίζονται από χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και αγανάκτηση προς την κοινωνία. Ας ψάξουμε λοιπόν την ρίζα του προβλήματος, το τι δεν πάει καλά στην κοινωνία. Και το λέω αυτό διότι πιστεύω πως η γνωμοδότησή μας δεν θα ε, πρέπει να είναι μακροσκελής. Πιστεύω πως πρέπει να συγκεντρωθούμε στα ουσιώδη, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν επί τόπου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εστιάσει σε στις ε, αιστείες των προβλημάτων. Και πιστεύω ότι η ηθική παιδεία είναι πολύ σημαντική. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε που υπάρχουν προβλήματα και σε καμία περίπτωση να μην αφήσουμε την αγανάκτηση να κατακυριεύσει αυτούς τους νέους επειδή δεν ξέρουν τι να κάνουν πρέπει να τους δείξουμε προοπτικές προοπτικές για την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας. Αυτή είναι η περίληψή μου και σίγουρα πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Σας ευχαριστώ. Είχαμε μια πολύ πλούσια συζήτηση. Δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς να παρέμβετε Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω δύο λόγια. Ο Επίτροπος στην πρόσφατη παρουσία του εδώ στην Επιτροπή παρουσίασε τη διακήρυξη του Παρισιού, την πρότασή του για την ασφάλεια και την ύψιστη προτεραιότητα για την Επιτροπή. Άκουσα πολύ προσεκτικά όλα όσα είπατε. Πρέπει να θυμάστε ότι και η διακήρυξη του Παρισιού αλλά και η ατζέντα για την ασφάλεια στοχεύουν την πρόληψη. Και φυσικά η εκπαίδευση πρέπει να και μπορεί να παίξει εδώ ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την πρόθεση των ε, κοινών ε, θεμελιωδών αξιών μας, αλλά και για την καταπολέμηση αυτής της ε, ριζοσπαστικοποίησης. Φυσικά και πρέπει η προσέγγιση μας να αφορά πολλούς τομείς, νέους, τον πολιτισμό, αλλά και τον αθλητισμό. Υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και φυσικά παρακολουθούμε τις διάφορες προτάσεις σας για δράση και αν μπορούμε να ξαναμιλήσουμε για τα θέματα αυτά και να ανταλλάξουμε απόψεις, με μεγάλη χαρά θα ήθελα επίσης να σας πω ότι προετοιμάζουμε και μία πρόταση, μια κοινή έκθεση Επιτροπής Συμβουλίου για τα θέματα αυτά. Το σχέδιο θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο και βεβαίως από τη στιγμή που θα δημοσιευθούν θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Εδώ βεβαίως ε, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και στο θέμα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης για να αποφύγουμε αυτήν την ε, ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Και βεβαίως προωθούμε αξίες όπως η πολυμορφία, ο σεβασμός τη διαφορετικότητας κοιτώντας και ποια είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να στηρίξουν αυτήν την ε, πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως έλεγα, είχαμε μία σημαντική και πλούσια συζήτηση. Α, όχι, Μήπως ήθελε ο εισηγητής να μιλήσει. Μάλιστα. Επιβεβαιώνω λοιπόν τις ημερομηνίε οι οποίες είναι εξή. Αύριο προθεσμία για τις τροπολογίες. 15 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε στην Επιτροπή Πολιτισμού. 12 Οκτωβρίου στη Λίμπε. Και εμείς θα έχουμε την ακρόαση στις 15 Οκτωβρίου. Και το οποίο θα είναι μια ευκαιρία να εμβαθύνουμε στα θέματα αυτά με τους ε, ειδικούς με τους εμπειρογνώμονες και έχω την εντύπωση ότι η υποστήριξη που δίνουμε στην Λίμπρε ακριβώς είναι μια θετική προσέγγιση του πώς η παιδεία είναι ένα μέσο μαζί με άλλες δραστηριότητες, τα αθλητικά, τα, οι δημιουργικές δραστηριότητες, οριζοντίως δηλαδή, ώστε να ενταχθούν καλύτερα είναι οι άνθρωποι στην κοινωνία, να επιτηρούμε και να παρακολουθούμε πολύ στενότερα και καλύτερα όλες αυτές τις προσπάθειες και η πρόληψη όπως είπε και ο συνάδελφος Μαραγκάλ είναι αν θέλετε μια επίπτωση δευτερογενής αλλά είναι αυτό που αποτυπώνουμε πολλές φορές ως μέτριο, μέτρο που μπορεί να αναλυφθεί. Να περάσουμε τώρα ευχαριστώντας όλους τους συμμετέχοντες την γνωμοδότηση του κυρίου Κρασνοντέτσκι για τις πολιτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων για την καταπολέμηση ενεργείας των νέων και για να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο συζήτηση και στις τροπολογίες μετακινήσαμε την ψηφοφορία στην ε, Επιτροπή Πολιτισμού στις 15 στην ΕΠΛ Έχουμε αναβάλει για 10 Νοεμβρίου, έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Και η προθεσμία υποβολής τροπολογιών 22 Ιουλίου. Δίνω λοιπόν το λόγο στο συνάδελφο Κρασνοντεύσκη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεδομένου ότι η συνεδρίασή μας θα κρατήσουμε το απόγευμα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ήδη ακούσαμε πολλά για το σοβαρό πρόβλημα τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων και ε, η γνωμοδότησή μου αφορά την καταπολέμηση της μεγάλης ανεργίας των νέων. Ενδεχομένως αυτά τα δύο συνδέονται. Φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι οι ε, αιτίες της ανεργίας ε, είναι διάφορες Ορισμένα στατιστικά στοιχεία ε, δείχνουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ε, είναι όπως θα έπρεπε, πως έχει κάποια προβλήματα. Από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχουν, υπάρχει μεγάλη ανεργία στους νέους, υπάρχουν όμως και πολλές κενές θέσεις εργασίας. Χρειάζεται να γεφυρώσουμε το το κενό. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να το αιτιολογήσουμε με το ότι οι δεξιότητες που έχουν οι ανεργηναίοι δεν είναι αυτές που ζητάει αγορά εργασίας. Η νέα γενιά όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε όλοι ότι είναι η γενιά με τις καλύτερες δεξιότητες. Ταυτόχρονα όμως είναι και η γενιά που μαστίζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη από την ανεργία. Εν κάνουμε μία αξιολόγηση όλων αυτών των στατιστικών στοιχείων θα ε, δούμε ότι αυτά προέρχονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία αξιολογούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο τους ε, μαθητές τους, φοιτητές τους, όμως αυτός ο τρόπος είναι διαφορετικός από εκείνον ε, τον οποίο χρησιμοποιεί η αγορά εργασία για να τους αξιολογήσει. Υπάρχει λοιπόν διαφορά αντιλήψεων και αυτό το πρόβλημα ε, πρέπει να επιλύσουμε. Τι προσπαθώ τώρα να κάνω με τη γνωμοδότησή μου. Θα αναφερθώ σύντομα σε ορισμένα ζητήματα και σε ορισμένους τρόπους που ενδεχομένως μας βοηθήσουν να κάνουμε την εκπαίδευση πιο αποτελεσματική έτσι ώστε να προετοιμάζονται οι νέοι άνθρωποι για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να βρουν γρήγορα δουλειά. Ε, αναφέρθηκε το επιτυχημένο μοντέλο του συστήματος διπλής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης ταυτόχρονα και σίγουρα είναι ένα σύστημα το οποίο, θα, το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. σε ενδεχόμενη εφαρμογή αυτού του συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα χρειαστεί ορισμένα κράτη-μέλη να ενισχύσουν την συνεργασία των ε, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τους ε, εργοδότες για διάφορα προγράμματα μαθητείας, για νέους, για φοιτητές, για μαθητευόμενους, να ενισχύσουν τα προγράμματα πρακτικής, διότι φυσικά όποιος ε, έχει στο τέλος των σπουδών του και ε, κάποια επαγγελματική εμπειρία θα είναι και πιο εύκολο να απορροφηθεί στην αγορά εργασίας. Χρειάζονται βέβαια κονδύλια για να στηριχθούν αυτά τα προγράμματα. Και Εάν δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, θα παρατηρήσουμε ότι νέοι οι οποίοι έχουν, τρίτο, έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν περισσότερες δεξιότητες και καλύτερες πιθανότητες να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας μετά το πέρας των σπουδών τους. Οι εκπαιδευτικοί έχουν επίσης πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Θέλουμε οι νέοι άνθρωποι να αποκτήσουν δεξιότητες και για να γίνει αυτό και για να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η εκπαιδευτική είναι πάρα πολύ σημαντική τα Ευρωπαϊκή Επιτροπή την χρήση των νέων τεχνολογιών, των ψηφιακών τεχνολογιών και εδώ πρέπει να αναφέρουμε τον ψηφιακό αποκλεισμό που ε, υπάρχει σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης. Η απόκτηση λοιπόν ψηφιακών δεξιοτήτων είναι κάτι που πρέπει να προωθείται στα σχολεία. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία που πρέπει να εξετάσουμε από τη μία λέμε ότι χρειάζεται καλύτερη σύνδεση ανάμεσα στην αγορά εργασίας, στην επαγγελματική κατάρτιση, και στην επαγγελματική κατάρτιση. Η επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να είναι ε, στοχευμένη στα επαγγέλματα που ε, παρουσιάζουν ε, μεγάλη ζήτηση. Και Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι δεν χρειάζεται μόνο εξειδίκευση, αλλά και γενικότερη κατάρτιση και, και καλύτερη παιδεία στις ε, ανθρωπιστικές επιστήμες. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ε, ψηφιακές ε, τεχνολογίες, τις νέες τεχνολογίες, αλλά να μην ξεχάσουμε και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τη λογοτεχνία, την κλασική παιδεία, την ε, εκπαίδευση στην ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά, τη μουσική. Χρειάζεται να μεταδώσουμε στους νέους ανθρώπους δεξιότητες οι οποίες θα καταπολεμήσουν τη ριζοσπαστικοποίηση. να εστιάσουμε στην παράδοσή μας, στην παραδοσιακή λογοτεχνία, την παραδοσιακή μουσική, διότι όπως είπα και πριν είναι καλή εξειδίκευση αλλά χρειάζεται και γενική παιδεία. Έχουμε παρατηρήσει επίσης φαινόμενα ανθρωπιστικής κρίσης σε ορισμένα κράτη-μέλη στον τομέα της, ε, στον τομέα της τέχνης, στην εκπαίδευση και χρειάζεται να εκπαιδευτούν οι νέοι άνθρωποι, να προσφέρουν τα σχολεία μαθήματα κλασικής παιδείας, ανθρωπιστικές επιστήμες. Από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τις, ε, τους τεχνίτες, διότι βλέπουμε μεν τα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων να είναι γεμάτα από φοιτητέ που σπουδάζουν πολιτικές επιστήμες, όμως ίσως θα ήταν καλύτερο ορισμένοι από αυτούς να ήξεραν ότι είναι προτιμότερη μια γενικότερη εκπαίδευση, ότι είναι προτιμότερο να μάθουν μια τέχνη και να εξειδικευτούν παρά αυτή η γενική παιδεία. Χρειάζεται η σωστή ισορροπία. Συμφωνώ με πάρα πολλές από τις ε, παρατηρήσεις σας, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Νέκοφ, δύο λεπτά ο καθένας σας παρακαλώ για να προλάβουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή για, το, για τη δουλειά σε αυτή τη χνομοδότηση. Η ανεργία των νέων είναι ένα κρισιμότατο πρόβλημα στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση η χρηματοπιστωτική και οι πολιτικές λιτότητες οδήγησαν αναπόφευκτα ε, στα επίπεδα ενεργείας των νέων που έχουμε αυτή τη στιγμή συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να, ε, να μετατρέψουμε τον τομέα της εκπαίδευσης ε, και την αγορά εργασίας ώστε να προσανατολίζεται με αμεσότερο τρόπο στη διοχέτευση των νέων ή στην αγορά εργασίας. Διαπιστώνουμε ότι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα ενημέρωσης και εκπαίδευσης αλλά αυτό είναι μόνο μία πτυχή του προβλήματος. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω έξι κρίσιμα στοιχεία σχετικά με το πρόβλημα αυτό. μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση των πρωτοβουλειών και των προγραμμάτων που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Προκειμένου να έχουμε μια βιώσιμη λύση πρέπει να έχουμε και έγκαιρα μέτρα θα πρέπει να έχουμε ένα διαφρομένο διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας και της αγοράς για να, για να τροποποιούμε τα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα προς τις ανάγκες της αγοράς. Θα πρέπει να αναπτύξουμε επίσης δεξιότητες ε, βάσης μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ε, προχωρημένες ε, δεξιότητες και τεχνική κατάρτιση στην ψηφιακή τεχνολογία, στα μαθηματικά ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ε, αυξημένες και συνεχώς μεταλλασσόμενες ανάγκες της αγοράς. Πρέπει να δούμε και τα επίπεδα μισθολογικής ε, προσέλκυσης των νέων, διότι αυτή τη στιγμή σχεδόν σε όλα τα επίπεδα της αγοράς συμπεριλαμβανομένων βασικών ε, σπουδών όπως ε, της μηχανικής ε, και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας δεν έχουμε θέσεις εργασίας με αρκετά υψηλές απολαβές. Εγώ θεωρώ ότι και τα συστήματα εκπαίδευσης ε, για τους μάνατζερ θα πρέπει να ενταχθούν και στην επίσημη και την άτυπη παιδεία και εκπαίδευση. Επίσης, σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό θα πρέπει να λάβουμε πάρα πολύ σημαντικά υπόψη μας το φαινόμενο της πρόορης εγκατάλειψης των σχολικών σπουδών μεταξύ των δεξιοτήτων βάσεως που σας ανέφερα νωρίτερα. Και για να βρούμε βιώσιμη λύση για την ενεργεία των νέων θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εγγυηθούν ε, επαρκή χρηματοδότηση προγραμμάτων υψηλής επαρκούς περιπτώσει ποιότητος. Οι επενδύσεις ε, στην παιδεία είναι πρώτη προτεραιότητα προκειμένου να έχουμε, να εξασφαλίσουμε ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε πρέπει να το κάνουμε μέσω της παιδείας, της παιδείας και ακόμα της παιδείας. Τρούπελ και μετά Ροϊντρόβα λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον ε, εισηγητή και θα ήθελα να πω ότι σίγουρα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να δώσουμε περισσότερε ευκαιρίε και περισσότερε δυνατότητε στους νέου ανθρώπου. Θα σταθώ όμω σε αυτά που είπε ο κύριο ε, Κρασνοδέψκη στο τέλο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η γενική παιδεία στι ανθρωπιστικέ επιστήμες και πόσο, ε, μπορεί, πόσο μπορεί να προσφέρει αυτή σε κάποιον νέο άνθρωπο και πώ μπορεί μέσω αυτών να αποφύγει τη ριζοσπαστικοποίηση. Ε, η παιδεία δεν είναι μόνο εξειδίκευση. Πρέπει να ε, δούμε την παιδεία ως σκοπό ε, αυτοεκπλήρωσης. Δεν, είναι, δεν πρέπει να είναι ο μοναδικός μας στόχος να δημιουργήσουμε καταρτισμένους ανθρώπους για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Πρέπει να δούμε ότι οι δεξιότητες αναπτύσσονται και μέσω των ε, ανθρωπιστικών σπουδών και μέσω των ε, επαφών ανάμεσα στις, στους πολιτισμούς μέσω ε, της εμβάθυνσης στην γενικότερη παιδεία. Τώρα όσον αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και σχετικά με το δικό σύστημα εκπαίδευσης. Ε, έχουμε την εμπειρία από πολλές ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη δική μου τη Γερμανία ε, ενός συστήματος που έχει αποτέλεσμα. Πρέπει όμως να προσέξουμε, να μην εξάγουμε αυτό καθ' αυτό ε, αυτούσιο το σύστημα στις άλλες χώρες, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να το προσαρμόσουμε στις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους. Εάν καταφέρουμε κάτι τέτοιο, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για επιτυχημένη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Χρειάζεται όμως προσοχή. Ευχαριστώ. Η κυρία ε, Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα να σας πω ότι θα ήθελα να προσθέσω κάποια στοιχεία σε αυτή την έκθεση. Καταρχήν συμφωνώ με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Πρέπει να επικεντρωθούμε στις δυνατότητες να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας αυτοί οι νέοι και βεβαίως θα πρέπει να μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα, κάτι που θα πρέπει να ενσωματώσουμε στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στα προγράμματα κατάρτισης, επιχειρηματικότητα λοιπόν που πρέπει σίγουρα να ενσωματωθεί στην έκθεση αυτή γιατί με αυτόν τον τρόπο οι νέοι θα μπορέσουν ευκολότερα να βρουν δουλειά. Δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα, ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός η σταδιοδρομία ενός νέου, ο επαγγελματικό του προσανατολισμός πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί, γιατί πολλές φορές υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό που ψάχνει ένας νέος και στις ανάγκες της αγοράς. Βλέπουμε ότι σήμερα 40% μιας ε, συγκεκριμένης ε, ομάδας νέων έχει πτυχία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι να είναι μία εκπαίδευση ποιότητας και κυρίως σε τομείς που αντιστοιχούν στις ανάγκες της αγοράς. Η επαγγελματική κατάρτιση και η εκπαίδευση που γίνεται εκ στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις επιχειρήσεις πρέπει επίσης να προωθηθεί. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν, λέει η Πρόεδρος, θα ήθελε να παρέμβει. Όχι. Άρα θα περάσουμε στην απάντηση του εισηγητή, εφόσον το επιθυμεί βεβαίω. Αλλά βλέπω γενική συμφωνία Θυμίζω ότι η προθεσμία είναι 22 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Και μετά θα ψηφιστεί στις ε, ενόψη της ακρόασης της 15ης Οκτωβρίου. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή γνωμοδότηση για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και θα μπορούσαμε να περάσουμε τώρα στην ε, γνωμοδότηση του κυρίου Μπαραντιαράν για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα Ηνωμένα Έθνη και την εξωτερική πολιτική, το οποίο εντάσσεται σε αυτήν την ε, νέα ερμηνεία της Επιτροπής Πολιτισμού να είναι πιο, πιο παρούσα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση για το ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη και κάποιες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής είναι ο, είναι ο τρόπος για να μιλήσουμε για μια πραγματική και πλήρη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο διαπολιτιστικός διάλογος. Ε, η ίδια η έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς αυτή η πολιτιστική διαφορετικότητα. Οι πολλαπλές ταυτότητες. Θεωρώ λοιπόν ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να είναι το κλειδί για την καλύτερη συνεννόηση και προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη διεθνή σκηνή όπως είναι η τρομοκρατία, όπως είναι οι μεταναστευτικές ροές πολιτιστική διπλωματία δεν σημαίνει απλώς να διοργανώνουμε μουσικές εκδηλώσεις. Σημαίνει να εστιαζόμαστε στις πολιτιστικές δραστηριότητες και αξίες και να εργαζόμαστε κατά τρόπον ώστε ο πολιτισμός να γίνεται soft power στις διπλωματικές μας επαφές και σχέσεις και προκειμένου να διαχέουμε τα δημοκρατικά ιδεώδη και τις δημοκρατικές αξίες που υποστηρίζουμε και να αναπτύσσουμε σχέσεις παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών. Οικοδόμηση δηλαδή γεφυρών σχετικά με την υποστήριξη των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπό την έννοια αυτή η συνεργασία μας με τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τα θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού και σημειώνω απλώς την UNESCO σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να χαρακτηρίζεται από καλύτερη εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής και πιο δραστήρια συμμετοχή σε συγκεκριμένες περιοχές όπως η προστασία της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς και των έργων τέχνης και όλα αυτά ως μέσο βιώσιμης ανάπτυξης ή την καλύτερη διαχείριση των ε, ε, στρατοπέδων προσφύγων σε διάφορες χώρες με πόλεμες ε, σειράξεις. Νομίζω ότι καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία που συμπεριλαμβάνει αρκετές στοιχείες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και τις αναφέρουμε στην, στο κείμενο, στην έκθεση αυτή. Εμείς ζητούμε από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσεως σε κάθε αποστολή στο εξωτερικό να υπάρχει ένας υπεύθυνος συντονισμού των πολιτιστικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινή δράση με τους εταίρους μας. Να προαγάγουμε την κινητικότητα των ε, δημιουργών, των καλλιτεχνών, δίδοντας συγκεκριμένα κίνητρα και βελτιωμένες συνθήκες, στο ίδιο πλαίσιο που χρησιμοποιεί και η UNESCO για την προώθηση των ε, ε, έργων τέχνης και των δημιουργών. Αυτή ακριβώς η σύμβαση την οποία προσυπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση και που γιορτάζουμε ακριβώς φέτος τα δέκατα γενέθλιά της είναι μια παρακολούθηση της παγκόσμιας διακήρυξης για την πολιτιστική ταυτότητα που ενεκρίθη μόνο λίγες εβδομάδες μετά από τα χτυπήματα της 11 η Σεπτεμβρίου του 2001 και εκεί μιλούμε για την πολιτιστική διαφορετικότητα ως ε, πεδίο δημιουργικότητας και αμοιβαίων ανταλλαγών που είναι απαραίτητο για την βιωσιμότητα των πολιτισμών σαν να ήταν ζώντες οργανισμοί. Εδώ μιλούμε για, τον, για το κοινό έδαφος καλλιέργειας της ανθρωπότητας του παγκόσμιου πολιτισμού και είναι απαραίτητο τόσο για τις τωρινές όσο και για τις μελλοντικέ γενναίες. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε σε τόσο δύσκολες στιγμές την απόλυτη αξία και χρησιμότητα του, διάλο, του διαλόγου, με συγχωρείτε, ώστε να μπορούμε να συνυπάρχουμε ειρηνικά ή τουλάχιστον να το προσπαθούμε. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Οι σκιώδεις τώρα ζήτησαν το λόγο, Στουργέτσκι, Ενέκοφ, Μπάσκι και Τρούπελ. E, Θα ήθελα να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ γρήγορη ανάγνωση αυτού του κειμένου. Λυπάμαι λοιπόν τους Γερμινείς. Τέλος πάντων, πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό και οι προτάσεις αυτές ε, είναι εξαιρετικά συγκεκριμένες. Τις υποστηρίζω λοιπόν. Το ίδιο και τις τροπολογίες. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω μία συγκεκριμένη πτυχή. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε δύο πτυχές. Ο πολιτισμός περιέχει ένα σύνολο αξιών. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τους δημιουργούς, τα έργα τους και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Υπάρχει όμως και μια άλλη διαδικασία που είναι η χρήση, η χρησιμοποίηση του πολιτισμού για να προωθήσουμε την ανάπτυξη των κοινωνιών μας στην Ευρώπη. Και αυτό σαφώς και προϋποθέτει διαφορετικά εργαλεία και μέσα. Για να προωθήσουμε έναν καλλιτέχνη χρησιμοποιούμε διαφορετικά μέσα από το όταν προσπαθούμε να προωθήσουμε τον ίδιο τον πολιτισμό. Και αυτό είναι κάτι που θα ήθελα οπωσδήποτε να το κάνουμε καθότι ο ΙΕ δίνει ιδιαίτερη σημασία στις διαδικασίες αυτές. изключително кратък. Имаше един Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει πολύ επικοδομητικός διάλογος με τον εισηγητή. Και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη συνεργασία μεταξύ του ΟΙΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία της ε, παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας. Το ίδιο θα έλεγα και για την προστασία της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς σε εμπόλεμες ζώνες. Μετά την ε, υπογραφή του μνημονίου η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και UNESCO βελτιώθηκε πολύ σημαντικά. Γι' αυτό και θα ήθελα να προτείνω μία ομάδα η οποία θα έχει σαν σκοπό να προωθήσει αυτό το διάλογο μεταξύ Ηνωμένων και Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε υψηλό επίπεδο έτσι ώστε να μην λειτουργούμε πάντα βάσει ενός κατεπήγοντος σχεδίου ή προγράμματος. Για να προστατεύσουμε καλύτερα την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά χρειάζεται λοιπόν ένας διαρθρωμένος διάλογος. Στα πλαίσια των συγκεκριμένων αυτών μέτρων πρέπει να στηρίξουμε τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες αυτούς που έχουν συγκεκριμένα σχέδια και τα οποία θέλουν να τα υποστηρίξουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαμπάσκη, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να υποστηρίξω τις τροπολογίες και τις προτάσεις που ακούστηκαν. Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο για να προετοιμάσουμε την έκθεση αυτή. Έχω υποβάλει τροπολογίες εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας. Το θέμα του καθεστώτος του παρατηρητή για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ηνωμένα Έθνη. Ο εισηγητής προτείνει να δώσει δικαίωμα ψήφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα για υπηρεσίες και φορείς που υπάρχει πολιτιστικό αντικείμενο. Δεν έχει νόημα σήμερα να ζητήσουμε δικαίωμα ψήφου αν δεν έχουμε δικαίωμα να υπερασπιστούμε τα πολιτιστικά προγράμματα τα οποία ε, προτείνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Η κυρία Τρούπελ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον συγγητή. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πολιτισμική έννοια στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών είναι μια πτυχή των εξωτερικών σχέσεων που πιστεύω πως ε, αφορά περισσότερο τις διαπολιτισμικές σχέσεις. Έχει να κάνει με το, με, τη, με το να δώσει περισσότερες δυνατότητες στους πολίτες να επικοινωνήσουν ένας με τον άλλον. Είναι ένα ζήτημα χειραφέτησης των πολιτών, αν θέλετε. Εγώ θα ήθελα να τονίσω πως χρειάζεται να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στους πολίτες και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με συνεργασία με τις αμή κυβερνητικές οργανώσεις, όχι μόνο με τα θεσμικά όργανα. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφής ο ρόλος μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε καλύτερα στα πλαίσια αυτού και να ενισχυθεί ο διάλογος με τους πολίτες. Επίσης, γίνεται πολλής λόγος για συγκρούσεις και πρέπει να αναφερθεί, πιστεύω, η ε, δυνατότητα αντιμετώπισης κρίσεων. Χρειάζεται επίσης τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Εάν δώσεις τους ε, ανθρώπους πολιτισμικές δυνατότητες ε, για να έρθει πιο κοντά ένα στον άλλο, τότε αυτό θα βοηθούσε πραγματικά. Και θα υποβάλω μια σχετική τροπολογία. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ούτε εδώ φαντάζομαι ότι η Κομισιόν κάτι θέλει να σχολιάσει. Λοιπόν, ο εισηγητής θα ήθελε να απαντήσει, να παρατηρήσει κάτι. Μόνο πολύ σύντομα, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Όπως και τους ε, σκιώδεις εισηγητές που τοποθετήθηκαν, είναι περίπλοκη η έκθεση. Προσπαθεί να καλύψει με λίγα λόγια αρκετά και περίπλοκα θέματα και για να καλύψει και να εντάξει τις ε, προτινόμενες τροπολογίες προς την Κομισιόν θα είχα το ξεκάθαρο αίτημα να μην παραδοθούμε και να προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε να έχουμε περισσότερη Ευρώπη ιδιαίτερα σε θέματα όπως αυτά που ανέφερα δηλαδή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε μια ακτίνα δράσεως όχι μόνο συγκρίσιμη με τις χώρες εταίρους αλλά για να συνεργαστούμε καλύτερα και με τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Εγώ προσωπικά θα πω ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψω ποτέ το ευρωπαϊκό ιδεώδες σε αυτό το επίπεδο της προσπάθειας σα ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το μήνυμα που δίνουμε της ενισχυμένης συνεργασίας ε, της πολιτιστικής, δηλαδή συνεργασίας στο πλαίσιο της εξωτερικής ιεραρχής πολιτικής, γιατί ίσως να είναι μια οδός ώστε να κατανοήσουμε από κοινού ή να κατανοήσουμε καλύτερα κάποιες από τις βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής ε, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετικότητα και χρησιμοποιώντας αυτήν τη soft power που αναφέρετε κι εσεί ω ε, πολιτιστική διπλωματία. Νομίζω ότι αυτή είναι επίση μια καλή ευκαιρία ώστε να εντάξουμε και το θέμα που εχθέ ε, συζητήσαμε. Δηλαδή, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, των έργων τέχνης, των μνημείων, την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου των αγαθών αυτών, αλλά και την αντιμετώπιση αυτών των εκτάκτων αναγκών με τα εκατομμύρια των προσφύγων που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, το θέμα του διαπολιτιστικού διαλόγου, που όλο και περισσότερο είναι ένα τμήμα, αν θέλετε, εξωτερικής πολιτικής και εν πάση περιπτώσει πολιτικής γειτονίας. Και επίσης εις τους στόχους της χιλιετίας. Γιατί νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν στην ακόλουθη σύνοδο της Άντις Αμπέμπα για τους στόχους της χιλιετίας και σε επικείμενη διακυβερνητική διάσκεψη που θα ασχολείται με το ζήτημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Στις 15 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία μας για τις τροπολογίες. 15 Οκτωβρίου ψήφιση στην Επιτροπή μας και στην ΑΦΕΤ 13 Οκτωβρίου. Έχουμε λοιπόν κάποιο χρόνο. Τι άλλο έχουμε. Α, ναι. 14 Σεπτεμβρίου στις 3 η ώρα είναι η επόμενη συνάντησή μας και 15 Σεπτεμβρίου σε 9 το πρωί. Να ευχαριστήσω τους ολίγους αλλά πανάξιους συναδέλφους που παρέμειναν μαζί μας και να ευχηθώ σε όλους πολύ καλές διακοπές. Να ευχαριστήσω τη γραμματεία, τους συμβούλους, τους policy advisor, τους βοηθούς, άπαντες. Σας ευχαριστώ που μείνατε ως το τέλος. Καλές διακοπές σε όλους. Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο.